Okay, colleagues, I'm going to begin um, Λοιπόν, ας αρχίσουμε συνάδελφοι. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε ξανά, μιλώ πάλι στα νέα μέλη, όταν αρχίζουμε αργά τη συνεδρίαση καταντάμε να κάνουμε αυτά που κάναμε χτες. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, συμπιέζουμε το χρόνο ομιλίας και ο καθένας θέλει να μιλήσει και καταλαβαίνετε μετά ζοριζόμαστε στο τέλος και θέλω πάντα να ξεκινάμε στην ώρα μας, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Για τα παλαιότερα μέλη και για τα νέα λέω ότι αυτό θα είναι το ύφος μου, αυτό με το οποίο θα προεδρεύω από την ώρα μας. Από το Σεπτέμβριο ακριβώς την ώρα θα αρχίζουμε. Κάτι άλλο πάλι για τα νέα μέλη. Μου είπαν ότι ε, θα θέλανε κάπως να τους εξηγήσουμε τις μυστήριες ε, μεθόδους ε, που ισχύουν εδώ μεταξύ αυτών και για τα κινητά αν είναι ανοιχτά κλειστά εγώ το σβήνω και το έχω ζεστό κατά τη διάρκεια ε, τις συνεδρίασης από το Σεπτέμβριο. Θα πούμε και κάποια διαδικαστικά που είναι δύσκολα για τον προϋπολογισμό και αυτά. Ακόμα και έμπειρος βουλευτής να είσαι καμιά φορά μπερδεύεσαι. Ε, προϊόντος του χρόνου θα ε, εξηγούμε διάφορα πράγματα και να απευθύνεστε παρακαλώ και στα παλαιότερα μέλη που τα γνωρίζουν. Ανακοινώσεις έχω μερικές. Έχουμε μερικές ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο για τη μετανάστευση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ε, προηγουμένως όμως να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Ε, είπα και χτες στα νέα μέλη ότι αυτές οι ανακοινώσεις ε, ε, είναι σημαντικές. Ε, πρόκειται για διορισμούς, διορισμούς εισηγητών. Συνήθως στην ε, αρχή της συνεδρίασης εγκρίνονται ε, αυτά, οπότε καλό θα είναι να έρχεστε νωρίς και να το γνωρίζετε. Αλλά αν είναι εδώ οι βοηθοί σας θα τα ακούσουν εκείνοι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, καταρχάς, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 229 του κανονισμού, έχει ξεκινήσει κάποια νομοθετική δουλειά στην προηγούμενη ε, κοινοβουλευτική ε, περίοδο και θα πρέπει να επανοριστούν οι ε, συγητές για τα σχέδια νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν, αν είναι ακόμα βουλευτές βεβαίως. Και οι ομάδες κρατούν τις εκθέσεις μελών που δεν έχουν επανεκλεγεί, που δεν είναι πλέον βουλευτές και θα πρέπει να ορίσουν νέους ηγητές το συντομότερο. Ε, σύμφωνα με αυτό λοιπόν το άρθρο του κανονισμού ορίζονται εξή. Η κυρία Μέτσολα του ΕΛΚ για την έκθεση συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνομοσπονδίας της Ελβετίας για τη συμμετοχή της στο ΕΑΣΟ, η κυρία Ενετβέλτ από τους Φιλελευθέρους για τη συμφωνία Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά και χειρισμό των PNR ε, για τον προϋπολογισμό του 2015. Η έκθεση δόθη στο ΕΛΚ και στον κύριο Στεσχόφσκι. Οι ε, συντονιστές συμφώνησαν ένα σύστημα εκπεριτροπής ορισμού ετησίως ενός εισηγητού. Ε, υπάρχει ενδεχομένως μία ομάδα εισηγητών και σχεδόν εισηγητών για να έχουμε καλύτερη εικόνα του προϋπολογισμού από τη ΛΥΜΠΕ. Η επόμενη ε, ομάδα που θα ορίσει εισηγητή για τον προπολογισμό είναι οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και ακολουθούν κατά σειρά η CRL, De Gue, Green, Πράσινη και η FDD. Και η τελευταία μου ανακοίνωση είναι το γλωσσικό καθεστώς. Αποφάσισαν οι συντονιστές σε περίπτωση που είναι περιορισμένες οι εγκαταστάσεις στην αίθουσα τι σημαίνει όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι διαδικαστικά και γραφειοκρατικά και ως την ορολογία. Ε, και γλωσσικό καθεστώ, σημαίνει πόσες γλώσσες έχουμε και ποια διερμηνία. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν πάντα τις ανάγκες των τακτικών αλλά και των αναπληρωματικών μελών. Και ε, ορισμένα από τα αναπληρωματικά μέλη ε, στην Επιτροπή μας είναι δραστήρια, λαμβάνουν φακέλους. Ε, όταν είναι μικρότερες οι αίθουσες, ε, στους συντονιστές θα συζητείτε αυτό το θέμα και θα το δηλώνουν στη γραμματεία για το γλωσσικό καθεστώς. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, ε, θεωρούνται εγκεκριμένες όλες αυτές οι ανακοινώσεις που σας έκανα. Ωραία, ας πέρασουμε στην ημέρηση. διάταξη αυτή καθ' αυτή. Όπως σας είπα, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για θέματα μετανάστευσης, το ένα για το Σέγγεν. Αρχίζουμε λοιπόν θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη παρουσίαση. Ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά για σας. Είναι η οδηγία σχετικά με την επιβολή κυρώσεων και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτή η οδηγία εγκρίθηκε στις 18 Ιουνίου του 2009, όχι φέτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωσή της στις 22 Μαΐου ενεστώτος έτους και τώρα θα μας παρουσιάσει την ανακοίνωση αυτή και θα ακολουθήσει συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Σμίτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως πριν περάσω στην ανακοίνωση να πω ε, κάποια γενικά πράγματα για να σας δώσω το υπόβαθρο ε, και για, αυτό το, για την οδηγία και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Συζητήθηκε χθε το θέμα της μετανάστευσης. Ε, ξέρετε ότι έρχονται πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί κανείς να βρει και παράνομη εργασία ε, όντας ένας μετανάστης δηλαδή που δεν έχει νόμιμα, δεν διαμένει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος όλων αυτών των ανθρώπων είναι να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και δυστυχώς πολλές φορές ε, πέφτουν θύματα ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται οικονομικά ανειδίκευτους ε, εργαζόμενους, ε, χαμηλά αμοιβόμενες εργασίες, ξενοδοχεία, καθαριότητα κτλ. Και γνωρίζουμε επίσης ότι πολλοί πέφτουν και στα χέρια διακινητών. Η οδηγία αυτή έχει μεταξύ άλλων λοιπόν το στόχο της καταπολέμησης όχι μόνο της ε, παράνομης εργασίας αλλά και της εμπορίας. Ξέρουμε ότι η αδήλωτη εργασία ουσιαστικά στερεί το κράτος από έσοδα και, από... και στον τομέα των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει να το δούμε συνολικά λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Στόχος είναι να βελτιώσουμε το μηχανισμό, τους μηχανισμούς ανείχνευσης, να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, με τους μετανάστες συγκεκριμένα, αν δεν έχουν πληρωθεί για τη δουλειά που έκαναν να πάρουν κάποια πληρωμή, κάποια στιγμή, κάποια αμοιβή. Φυσικά ότι και αυτή δεν στρέφεται κατά των μεταναστών, αλλά κατά των εργοδοτών που τους εκμεταλλεύονται. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι είναι συμπληρωματική προς μια πολύ πρόσφατη οδηγία η οποία λίγο πολύ καλύπτει τους ίδιους τομείς που καλύπτει η οδηγία που συζητούμε σήμερα, δηλαδή μιλώ για την οδηγία περί εποχικών εργαζομένων Η οδηγία για τους εποχικούς εργαζομένους άνοιξε κάποιες νομικές οδούς για τους εργαζομένους που αναζητούν νόμιμη απασχόληση. Εκδώσαμε λοιπόν τον Μάιο μία ανακοίνωση. Σε αυτήν τρεις βασικές προκλήσεις αναφέρονται σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Η πρώτη πρόκληση είναι η ανάγκη διενέργειας παρκού αριθμού επιθεωρήσεων στα κράτη-μέλη εάν αυτά δεν διαθέτουν ε, κατάλληλους μηχανισμούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιθεώρησης δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και την αντίλωτη εργασία, την παράνομη εργασία, ούτε μπορούν ε, οι μετανάστες ε, να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε αποτελεσματικούς ελέγχους τώρα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο Άπαξε ετησίως θα πρέπει να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη για τον αριθμό των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει, που εντόπισαν δυσκολίες, σε ποιους τομείς. Το 2013 πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση δεν ήταν και τόσο καλή. Δεν έδωσαν όλα τα κράτη-μέλη εκθέσεις. Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες παραβάσεις. Τέλος πάντων, ε, ε, λάβαμε όλες τις εκθέσεις και αναφορές για το 2012 που δείχνουν ότι οι τομείς που πλήγονται ιδιαίτερα από την παράνομη εργασία είναι οι ίδιοι σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή οικοδομή, γεωργία, ε, καθαριότητα, catering, ε, υπηρεσίες, ε, φιλοξενίες κτλ ξενοδοχεία. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους είχαμε διαφορές. Ένα ε, λιγότερο του ενός ε, σε κάποια κράτη ελέγχθηκαν, ενώ σε άλλες είχαμε φτάσει και σε ποσοστό 29% των εργοδοτών που ελέγχθηκαν. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην προσπάθεια επιβολής ε, στα κρατημέλη, άρα οι εργοδότες ε, που παραβαίνουν την νομοθεσία πολλές φορές ε, αποφεύγουν τη σύλληψη ή τη δίωξη σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Έχουμε τώρα ετοιμάσει ένα νέο δείγμα για τις θεωρήσεις αυτές. Είναι πολύ καλύτερη φέτος η κατάσταση Έχουμε λάβει μέχρι στιγμής όλες τις εκθέσεις από όλα τα κράτη-μέλη και αναλύουμε την κατάσταση που εν γέννη φαίνεται να έχει βελτιωθεί αισθητά. Παραλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντική η έλεγχη επιθεωρήσεις για την ανείχνευση της παράνομης εργασίας. Δεύτερη πρόκληση. Η πρόκληση αυτή σχετίζεται με το επίπεδο οικονομικών, διοικητικών, ποινικών κυρώσεων που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη απαγορεύουν ε, την απασχόληση λαθρομεταναστών, επιβάλλουν κυρώσεις, είναι σαφές αυτό, όμως οι κυρώσεις, ο βαθμός της σοβαρότητας της κύρωσης ποικίλει από το ένα κρατός μέλος στο άλλο, για παράδειγμα. Σε 16 κράτη-μέλη το πρόστιμο, το ποσό του προστίμου αυξάνεται αναλογικά. Από 300 σε ένα κράτος μέλος μπορεί να φτάνει τα 10.000 ευρώ σε ένα άλλο. Μεγάλες διακυμάνσεις έχουμε δηλαδή. Επίσης τα κράτη-μέλη έχουν ορίσει και ένα μέγιστο πρόστιμο σε άλλα κράτη-μέλη είναι 850 ευρώ, σε άλλα 100.000. Στα κράτη-μέλη, ή μάλλον ε, στα κράτη-μέλη πολλές φορές ο δικαστής είναι αυτός που θα επιδικάσει το πρόστιμο βλέπουμε και διακοιμάνσεις και εδώ. 500 και μέχρι και 500.000. Σε, σε κάποια κρατημέλη είχαμε μέχρι και 500.000 πρόστιμο. Αυτό είναι το ανώτατο. Εμείς εργαζόμαστε με τα κρατη για να υπάρξει μια συνεκτικότητα, μια ομοιογένεια κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των κυρώσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι οι ίδιες οι κυρώσεις όλα τα κράτη-μέλη, γιατί διαφέρει η οικονομική κατάσταση, το επίπεδο των αμοιβών, από το ένα κράτος μέλος αλλά Τέλος πάντων κάποια συνεκτικότητα πρέπει να υπάρχει και βέβαια ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ε, δαναστών, μια άλλη πρόκληση πολύ σημαντική, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, διευκόλυνση ε, των καταγγελιών ε, για να εφαρμοστούν προστατευτικά μέτρα για να επανορθωθεί η αδικία ε, την οποία υπέστησαν οι λαφομετανάστες. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν την κατάσταση με τα κράτη-μέλη. Λίγα είναι αυτά τα οποία έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο ε, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ε, για μη καταβληθείς αμοιβή, Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες ακόμη τους επόμενους μήνες. Ένα άλλο σημείο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνται συστηματικά οι εργαζόμενοι για τα δικαιώματά τους. Το προβλέπει ρητά η οδηγία, δεν έχουν όμως όλα τα κράτη-μέλη τέτοιες διατάξεις. Και τέλος, έλλειψη ενίοτε μηχανισμών σε κάποια κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και οι δυσκολίες ε, που προκύπτουν από τη λαθρομετανάστευση. Πάντα σε σχέση με τα δικαιώματα. Βλέπω λοιπόν, ε, μάλλον βλέπουμε ότι πρόκειται για μια οδηγία σημαντική, καινούρια ε, ακόμη σχετικά είναι. Οι προτεραιότητές μας για τους επόμενους μήνες είναι πρώτον η ενδελεχής εξέταση της μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κάτι το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε εντοπίσει ελλείψεις στις εκθέσεις και όπως είπα τώρα θα δούμε πιο αναλυτικά την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Έχουμε και διμερείς ε, συναντήσεις στα κράτη-μέλη και η ομάδα επαφή έρχεται σε, ε, συναντάται με όλους τους ειδικού για την ε, διευκρίνηση ζητημάτων που είναι ανοιχτά προς ερμηνεία. Αν οι διμερείς συναντήσεις, ή άτυπες επαφές δεν αποδώσουν, ξεκινάν, ξεκινάμε επίσημα διαδικασίες επί παραβάση, αν δεν εφαρμοστούν δηλαδή οι νέες διατάξεις, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στα κράτη-μέλη διορθώσεις. Και πάντα σε σχέση και με την οδηγία περικυρώσεων, επαναλαμβάνω ότι είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Η οδηγία είναι πολύ σημαντική. Οι μηχανισμοί εντοπισμού ανείχνευσης βλέπουμε ότι τουλάχιστον έχουν βελτιωθεί. αλλά εξακολουθεί, όπως είπα, ε, να χρειάζεται να γίνει κάποια δουλειά. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σμιτ. Να δώσω κάποιες βασικές οδηγίες για τη συζήτηση, κυρίως για τους νέους συναδέλφους, αλλά πολλοί ήταν ήδη εδώ χθες, από πρακτικής άποψης. εφόσον ε, την ώρα που κάνει την ε, παρουσίαση τη Επιτροπή παρακαλώ να ζητάτε το λόγο, ε, μπορείτε να σκόρετε το χέρι σα να ενημερώνετε την γραμματεία, Ω προ την συζήτηση. Βλέπετε ότι έχουμε τρει ανακοινώσει. Αυτό που θα γίνει δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε με του συζητητέ και το καθεξή. Είναι μια πρώτη συζήτηση με του συντονιστέ, αλλά είναι μια πρώτη συζήτηση αυτή. Οπότε μπορείτε να θέσετε τι ερωτήσει σα, να λάβετε το λόγο και μετά θα λάβετε και απαντήσει. Μετά, ε, έτσι καλώς είδαμε την ε, σχετική συζήτηση για την ε, ομάδα δράσης στην Μεσόγειο χθε. Και είδατε, το είχαμε συζητήσει και με τους συντονιστές, αποφασίστηκε να γίνει ενδεχομένως έρευνα ή ακρόαση για την ομάδα δράσης για τη Μεσόγειο. Μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους επιλογές ούτως ή άλλως, αλλά όταν κάνετε τα σχόλιά σας να θυμάστε αυτά τα διαφορετικά ζητήματα. Έχουμε την μπλε κάρτα, τις κυρώσεις και το σύστημα επαλήθευσης. Θα πρέπει να τα έχετε αυτά κατά νου. Το λέω λοιπόν ευθύ εξ αρχής για να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτές οι συζητήσεις. Το λόγο έχει ζητήσει Κυρία Σίπελ, Μπεργίτε, ευχαριστώ πρόεδρε. Στα αγγλικά. Καταρχάς θέλω να πω ότι χαίρομαι που στην οδηγία αυτή δεν μιλούμε μόνο για κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες, αλλά και για υποστήριξη στους ε, μετανάστες αν δεν έχουν πληρωθεί, αν έχουν κακοπληρωθεί από την άλλη, ενοχλούμε πολύ που ακούω ότι αυτή η οδηγία σε πολλά από τα κράτη-μέλη μας δεν βρίσκει συγκεκριμένη εφαρμογή, ούτε αποτέλεσμα, διότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ακούσαμε μεταξύ 1 και 29%, δηλαδή υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι μπορούν να αλωνίζουν και είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθούν. Και βέβαια οι ίδιοι έλεγχοι κοστίζουν. Και από την άλλη, όπως μας είπε η συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να γίνουν πολλές οικονομίες, διότι δεν καταβάλουν εργοδοτικές εισφορές, δεν πληρώνουν φόρους, ε, άρα τους συμφέρει τους εργοδότες. Εμείς θα πρέπει να ελέγχουμε τους εργοδότες. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εργάζονται ε, άνθρωποι που ζουν παράνομα στη χώρα, αλλά εργάζονται για μισθούς πείνας ε, σε πάρα πολύ κακές συνθήκες, δεν είναι ασφαλισμένοι και άλλα ε, πράγματα στερούνται. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η πολύ συγκεκριμένη μου ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι... Υπάρχει καμιά πιθανότητα κατά τη γνώμη σας να βελτιωθεί η κατάσταση στα κράτη-μέλη και να ε, τα αναγκάσουμε ή να τα ενθαρρύνουμε να κάνουμε περισσότερους ελέγχους για να βελτιωθεί η κατάσταση και για τους μετανάστες αλλά και για τους πάντες που ε, παρανομεί ή εργάζεται παράνομα ε, κανείς. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Θέλω να δω λιγάκι μαζί σας τα συμπεράσματα στο τέλος των γραφών σας, στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης λέγεται ότι το νομοθέτημα αυτό θα πρέπει να δώσει κίνητρα για να χρησιμοποιούνται νόμιμοι διαβλή για την μετανάστευση. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς εδώ, γιατί νόμιμοι διαβλή ακριβώ δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα ώστε να έχουμε ψηλή ε, παιδεία ε, μετανάστες και όχι μόνο του χαμηλότερη εκπαίδευση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί δραστικά και ο όγκος της μετανάστευσης προς ε, εμάς. Έτσι κι αλλιώς σε εμά έχουμε ελάχιστους ελέγχους στη χώρα μας, 1% σε σχέση με τους υπόλοιπους. Εάν λοιπόν αυξηθεί η νόμιμη μετανάστευση, δεν χρειάζονται και τόσες πολλές επιθεωρήσεις, τόση έλεγχη για ανθρώπους που είναι νόμιμοι. Έχουμε βεβαίω και κάποια προβλήματα, διότι κάποιοι εργοδότε είναι αδίστακτοι και πραγματικά εκμεταλλεύονται του εργαζομένου, αλλά θα πρέπει να ανατρέχουμε στην ισχύουσα νομοθεσία. Και δεν νομίζω ότι αρκεί να προβλέπουμε άδειε παραμονής για, τις για τους υψηλής μόρφωση μετανάστες ή του εποχιακού εργαζομένους. Πρέπει απλώς να έχουμε ένα σύστημα με μόνιμους και διαρκείς νόμιμους διάβλους για την μετανάστευση. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που απασχολούν λαθρομετανάστες κάποιες φορές δεν είναι αναγκαστικά ε, ανήθικοι. Απλώς μπορεί να πρόκειται για εθελοντικές οργανώσεις, για ιδιώτες που θέλουν να βοηθήσουν μονομένα άτομα που δεν έχουν κάποια δυνατότητα διαφορετική για να μείνουν σε μια χώρα ή να κερδίσουν τη ζωή τους δεν πρόκειται μόνο για ανθρώπους ε, σατανικούς που έχουν σκοπό να εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μελινέρ. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you, uh, Chair, for... Ευχαριστώ. Δεν σας άκουσα. Ε, ευχαριστώ και την κυρία Σμιτ που ήρθε σήμερα εδώ και μας έκανε αυτήν την διεξοδική παρουσίαση για, μια τόσο κρίσιμη, για ένα τόσο κρίσιμο θέμα για να δούμε τις ελλείψεις αυτής της οδηγίας. Δεν θέλω να μπω στις οδηγίες, τα, ε, παρουσιάσατε τα προβλήματα των αποκλήσεων μεταξύ ε, των κρατών μελών προς την υλοποίηση αυτής της οδηγίας, τις οικονομικές και ποινικές κυρώσεις. Τα συμπεράσματα τη ε, ανακοίνωση είναι πραγματικά ανησυχητικά, όπω είπατε και εσεί οι δύο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν θα προταθεί τροποποίηση τη οδηγία. Η δική μου λοιπόν σύσταση προς εσάς, ερώτηση προ εσά είναι πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βεβαιωθεί ότι το ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίηση τη οδηγία επιτυγχάνεται ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσει μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να ε, συνταχθούν κατευθυντήριες ε, γραμμές για την ε, πρακτική υλοποίηση της οδηγίας μεταξύ άλλων και της επιβολής των δικαιωμάτων των μεταναστών και των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση τέτοιων κατευθυντηρίων γραμμών. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σατόφσκι. Θα μιλήσω τσεχικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και την κυρία Σμιτ για την παρουσίασή της. Μία ερώτηση θα είχα μόνο. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε λίγο παραπάνω σχετικά με τους ελέγχους. Κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες θα με ενδιαφέραν και ιδιαίτερα ποιος διενεργεί ελέγχους και τι έλεγχοι είναι αυτοί και με ποιο τρόπο γίνονται. Διότι πιστεύω ότι αυτά τα ποσοστά δεν λένε και πολλά πράγματα. Μας λέτε από 1% μέχρι 29%. Ωραία, αλλά αυτό πώς αναλύεται, τι επιπτώσεις έχει και τι αντίκτυπο. Πριν εκλεγώ Ευρωβουλευτής, επί σειρά ετών ήμουν και εργοδότης. Δίφθηνα μια εταιρεία και ο αριθμός των ελέγχων είναι τέτοιος που δεν βοηθάει στο να αποκαλυφθεί αν κάποιος απασχολείται νόμιμα ή παράνομα ή αν είναι λαθρομετανάστης ή διαμένει νόμιμα. Παρακαλώ μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερα στοιχεία. Uh, Mrs. Bjork. Η κυρία Bjork. Okay. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας ενωτικής ε, αριστεράς και βόρειας πράσινης αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η νομική βάση και το υπόβαθρο αυτής της οδηγίας. Υποτίθεται ότι ο στόχος είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ε, σύμφωνα με την κεφαλίδα, ας πούμε. Χαίρομαι που ενισχύουμε τα δικαιώματα των μεταναστών στην οδηγία. Όταν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομιλεί για τις διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, το πρόβλημα είναι ακριβώς ένα ζήτημα δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ήρθαμε σε επαφή με πολλές οργανώσεις που εργάζονται και βοηθούν ανθρώπους σε αντίστοιχη κατάσταση και μας λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Πρώτον, να τιμωρηθεί στη συνέχεια από τον εργοδότη σου, γιατί εκτίθεσε σε διαφόρους κινδύνους, μέχρι και φυλάκιση ή και απέλαση και επίσης μπορεί κάποιος να ε, βρεθεί στη θέση που θα τον καταδώσει ο ίδιος του εργοδότης. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτών των εργαζομένων να διεκδικήσουν ε, μισθούς που τους οφείλουν και δεν τους έχουν καταβάλει. Και τελικά γίνονται και θύματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα μεταναστών που δεν έχουν χαρτιά. Όταν μιλάμε για περισσότερους ελέγχους και περισσότερες κυρώσεις, ίσως να μην είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτός να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα ήταν αποτελεσματικότερο ενδεχομένως να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, να είναι σε θέση να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους και να καταγγέλουν εκείνοι τους εργοδότες που τους εκμεταλλεύονται. Και θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για αυτό το τελευταίο, ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Stevens. Ja, Nu... Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίε, Έχω μερικές ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στους μετανάστες για να τους ενημερώσει. Εσείς πώς μπορείτε να φτάσετε ακριβώς για να τους ενημερώνετε για τα δικαιώματά τους, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται και με τις εργοδοτικές ε, οργανώσεις για να ευιστοποιούνται οι εργοδότες. Για να μην εργάζονται παράνομα ε, και στην μαύρη αδήλωτη εργασία, αλλά να ε, καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο μαζί με τους εργοδότες. Το ίδιο ισχύει και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. Μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και τα συνδικάτα ε, συμμετέχουν στη δική σας προσπάθεια. Ε, μπορούν να καταγγείλουν κάποιες καταστάσεις και κάποια κοσκήμενα ε, στην επιθεώρηση εργασίας, ακόμα και στην αστυνομία την ίδια. Οι εργαζόμενοι ε, των τρίτων ε, ε, χωρών είναι αυτό που μας ενδιαφέρουν, αλλά έχετε αριθμητικά στοιχεία και για εργαζομένους που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλη χώρα της Ένωσης και εργάζονται παράνομα σε μια άλλη χώρα μέλος. Δεν πρόκειται μόνο για επικόους τρίτων χωρών στο Βέλγιο. Έχουμε πολλούς ανατολικοευρωπαίους που έρχονται να εργαστούν σε αδήλωτη εργασία και ε, είναι ανασφαλιστή γιατί δεν καταβάλλονται ε, ασφαλιστικές τους εισφορές και τα ίδια ισχύουν για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία. Έχετε αριθμητικά στοιχεία να μας δώσετε. Επίσης, η ανακοίνωση λέει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Είναι πρόθυμες όμως αυτές οι τρίτες χώρες να συνεργαστούν. Μπορείτε να μας ενημερώσετε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Και επίσης, έχετε, ξέρω ότι είναι δύσκολη η ερώτηση, ποια είναι τα κράτη-μέλη που έχουν καλές επιδόσεις και ποιες είναι οι χώρες εκείνες που υπολείπονται. Ε, μιλήσατε για βέλτιστες πρακτικές. Έχετε κάνει κάποια αξιολόγηση εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω τι γίνεται με τη συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Εκεί ήδη υπάρχουν κάποιες κινήσεις, τις συζητήσαμε χθες το απόγευμα και στην Επιτροπή Απασχόλησης, μια πλατφόρμα ώστε να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη στα θέματα επιθεώρησης της αγοράς εργασίας, λόγου χάρη. Εξετάσαμε το θέμα αυτό εν μέρη, διότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αλλά και κάποια άλλα από αυτά που έφυξαν οι συνάδελφοι το πρωί, όπως τι γίνεται με την μεταχείριση των Ευρωπαίων επικών ή με τους εργαζομένους γενικότερα και τα δικαιώματά τους. Όταν η οδηγία αυτή εκρίθηκε, μία από τις ανησυχίες των εργοδοτών και για την απασχόληση είναι ότι οι έλεγχοι για τη μετανάστευση δεν θα πρέπει να μπερδεύονται με τους ελέγχους που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια στην εργασία λόγου χάρη. Δεν θέλαμε να παρεμποδίσουμε την πραγματική ε, υλοποίηση κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λόγου χάρη. Άλλα θέματα, ε, ανακατεύοντας δύο διαφορετικούς τομείς. Νομίζω τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αφορά όλους. Για κάθε όποια και είναι η προέλευση ενός εργαζομένου, είτε είναι μετανάστης, είτε Ευρωπαίος υπήκος και εδώ θα πρέπει να ενισχυθούν ε, τα σχετικά μέτρα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις πολιτικές της Τρόικας που ενδεχομένως να υποβαθμίζουν αυτά τα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Υπάρχει επίσης εδώ και μια διελκυστίνδα με το Συμβούλιο για θύματα που έχουν να κάνουν με την διεκδίκηση οφειλωμένων ε, αμοιβών. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα κάτι μέλη μπορούν να κατοχυρώσουν ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι απλώς να είναι μια διαδικασία αστική αυτή ώστε να ζητά κανείς τι αμοιβέ που το οφείλονται. Τι θα γίνει με έναν μετανάστη που έχει απελαθεί λόγου χάρη και τελικά δεν μπορεί να προσέλθει σε κάποιο δικαστήριο για να διεκδικήσει τι ε, οφειλόμενε αμοιβέ. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι έτοιμα να διαχειριστούν τα ζητήματα. Θα ήθελα απλώ σε πρώτη φάση να ακούσω όμω ποια είναι η διασύνδεση των ε, συζητήσεων σε εξέλιξη ε, που υπάρχουν ήδη στη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Υπάρχουν εκεί κάποιες κινήσεις που αν μη τι άλλο στα θέματα συνεργασίας ε, για την επιθεώρηση της αγοράς εργασίας θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρόεδρος. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε την οδηγία για του εποχικού εργαζομένους. Το μόνο υπάρχον νομοθέτημα για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να τα σκεφτούν αυτά, γιατί είναι πολλέ οι επιτροπέ που ασχολούνται με θέματα μετανάστευση, το καθεστώ των κυρώσεων στην οδηγία αυτή, τα ζητήματα τη ε, εργασιακή αγορά. Είναι πολλά τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας και μετά τη θέση σε σχέση της ε, συνθήκης. Υπάρχει λοιπόν εδώ και μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και εμείς συνεργαζόμαστε συστηματικά μαζί τους. Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι μέλη και σε εκείνη την Επιτροπή. Και αυτό εξηγεί και γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ και με θέματα μετανάστευσης, επιθεωρήσεων της αγοράς, της αγοράς εργασίας, τα δικαιώματα των μεταναστών και εργαζομένων και το καθεξής. Είναι ευαίσθητο θέμα των κυρώσεων. Οπότε θα μπορούσατε να δείτε και κάποιες πρώτες θέσει μας από τους τρεμερούς διαλόγους και ούτω καθεξής. Επόμενος. Ο μιλητής, η κυρία Weinberg ή Woodberg. Μπορείτε να μου πείτε τη σωστή προφορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την ε, ανακοίνωσή της αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Το ζήτημα αυτό και την εξέλιξή του θα τα παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή. Ήθελα απλώ να ακούσω λίγο περισσότερα για το πώς θα διεξαγάγονται ότι οι έλεγχοι. Είμαι νέα εδώ στο Κοινοβούλιο, νέα βουλευτής. Θα πρέπει να μελετήσω και εγώ το θέμα αυτό, αλλά ως προς τους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά στις επιδόσεις μας ε, για να γνωρίζουμε και πόσους ακριβώς ε, μετανάστες έχουμε στη χώρα, λαθρομετανάστες μάλλον. Προβλέπεται ελεύθερη υγειονομική περίθαλψη, ε, δωρεάν μάλλον υγειονομική περίθαλψη, ένα σωρό δικαιώματα για τους μετανάστες Οπότε, είναι ένα θέμα η έλεγχη. Τι γίνεται με τους μη ασφαλισμένους, τι γίνεται με αυτούς που μπορεί να τραυματιστούν ε, σε κάποια τύχημα και να πρέπει να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Παρακολουθούμε λοιπόν το ζήτημα με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το θέμα το βρίσκω πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι ε, το... εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε από τους χειρότερους μαθητές. Πρόεδρος, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των αγορητών είναι στη θέση της και η Προεδρία. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σύντομο σχόλιο, δεδομένου ότι είχαμε και τη συζήτηση για την ομάδα δράσης χθες, και μετά να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Βεβαίω και πρώτα απ' όλα με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα να βεβαιώσω και από την πλευρά μα την ιδιαίτερη προσοχή που θα δώσουμε στα θέματα τη μετανάστευση. Κάτι που θα μας απασχολήσει σε όλη τη διάρκεια της Αταλικής Προεδρίας και με διάφορες εκδηλώσεις που θα στρέφονται γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων των μεταναστών αλλά και των κυρώσεων. για την ε, οδηγία για τους ερευνητές, φοιτητές θα δείτε ήδη πώς η προσοχή και τις σχετικές συζητήσεις από αυτό το στοιχείο και μόνο βλέπετε η προσοχή δίνει η Προεδρία μας στο θέμα αυτό και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της συζήτησης για το θέμα που ε, ε η ανακοίνωση της Επιτροπής με ιδιαίτερη προσοχή. Πρόεδρος. Θα δούμε ε, εφόσον χρειαστεί, αν μπορούμε να οργανώσουμε και κάποια κρόαση, κάποια ομάδα ε, θα δούμε τι μπορεί να κάνει και από την πλευρά τη Προεδρία η Επιτροπή τώρα. Θέλετε να σχολιάσετε και να απαντήσετε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, όπως νομίζω αναφέρατε και εσείς ο ίδιος αλλά και κάποιοι βουλευτές, πρέπει να ακολουθήσουμε μια συνολική προσέγγιση και ακριβώς σε αυτή τη συνολική προσέγγιση εντάσσεται και η παρούσα οδηγία. Πρέπει να ανοίξουμε νομικές οδούς, ε, νομικούς διάβλους, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε μέσα στη διάθεσή μας, έχουμε τις οδηγίες ε, για τους υποχικούς εργαζομένους, για την οικογενειακή επανένωση όσων δεν έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες. Ε, μπλε κάρτα είναι ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια, οδηγία για τους φοιτητέ και τους ερευνητέ. Νομίζω λοιπόν ε, ότι καλό θα ήταν να έχουμε ένα φιλόδοξο κείμενο ώστε να ενθαρρύνουμε νέους ανθρώπους να έρθουν στην Ευρώπη μέσω νομίμων οδών. Και όλες αυτές τις οδηγίες ε, τις ε, εφαρμόζουν πλέον στο Εθνικό Δίκαιο τα κράτη-μέλη και δίνουν κάποια ευκαιρίες και κάποια δικαιώματα στους νέους. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι τα πάντα ε, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, πολλά είναι εθνική αρμοδιότητα. Να πω και στα κράτη λοιπόν να, ορίσουν κάποια ποσοστά, ποσοστώσεις για όσους έρχονται ε, στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη οδηγία αντιμετωπίζει την ε, λάθρο μετανάστευση, μεταξύ άλλων. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το λεγόμενο pull factor. Τη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων είναι ένα θέμα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις πίσω από τους ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές φέρνουν τους ε, μετανάστες σε επαφή με τους ε, εργοδότες που θα τους απασχολήσουν στη συνέχεια παράνομα. Άρα και αυτές οι πτυχές μας απασχολούν. Η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι επίσης σημαντική. Και τώρα θα ήθελα να επανέλθω στα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Σε σχέση με τις επιθεωρήσεις, να σας πω ότι προς το παρόν είναι νωρίς να πούμε αν βελτιώθηκε ή όχι η κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρώτη μας εντύπωση είναι ότι διενεργήθηκαν περισσότεροι έλεγχοι ή τέλος πάντων ε, είναι πληρέστερες οι πληροφορίες που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της ανάλυσης. Η οδηγία προβλέπει το ενδεχόμενο καθορισμού στόχων για τους έλεγχους, για τις επιθεωρήσεις. Το εξετάζουμε, θα δούμε αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο πώς μπορούμε να καθορίσουμε στόχους για τα κράτη-μέλη σε σχέση με την επιθεώρηση των εργοδοτών, λαμβάνοντας υπόψη και τους παρανόμως διαμένοντες εργαζομένους στα κράτη-μέλη. Δεν είναι η ίδια κατάσταση για όλα τα κράτη-μέλη, το τονίζω πάλι αυτό. Τέθηκε το ζήτημα της ενημέρωσης, είναι σημαντικό αυτό. Αν οι μετανάστες δεν είναι ενημερωμένοι, Εδώ μιλάμε για μια κατηγορία ανθρώπων στους οποίους είναι δύσκολο να παράσχει κανείς ενημέρωση λόγω της, ε, του νομικού καθεστώτος τους, ας πούμε, της νομικής τους κατάστασης. Σωστά υπόθηκε πάντως ότι πρέπει να ενημερώνονται. Επίσης και οι εργοδοτικές οργανώσεις πρέπει να ενημερώνονται για το μέλλον ε, δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων συζητήθηκαν αυτά τα θέματα και στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο και δεν υπάρχει μόνο η πτυχή της λαθρομετανάστευσης. Πρέπει και με τις επιχειρήσεις και με τα συνδικάτα και με τις εργοδοτικές ε, οργανώσεις να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και επαφή. Είχαμε επαφή με τους ε, φορείς αυτούς και στόχος μας είναι να δούμε αν μπορούν να διενεργήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο σε επίπεδο κράτους μέλους. Να μην ε, τα αφήνουμε μόνο δηλαδή στις αρχές των κρατών μελών. Το δικαίωμα κατάθεσης αγωγής, μήνυσης είναι ένα θέμα. Εμείς δεν θα διστάσουμε να κινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση, εάν αυτό χρειαστεί. Πάλι και εδώ είναι απαραίτητο να έχουμε την ενημέρωση. Τώρα για αυτή την πλατφόρμα γάμα απασχόληση, αυτό προτείνει Κομισιόν σε σχέση με την επιθεωρήση στην αγορά εργασίας. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τη γάμα δελτα απασχόληση όχι μόνο για το θέμα αυτό, γενικώ όλα τα ζητήματα που αφορούν την νόμη δικαιώματα λοιπά, όλα αυτά τα εξετάζουμε, παρακολουθούμε και τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο και μελετούμε και τις προτάσεις της, της ε, Γενικής Απασχόλησης. Ελπίζω να κάλυψα ε, τα μέλη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την κυρία Σμιτ. Είμαστε εντός χρονοδιάγραμμα, χρονοδιαγράμματος μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μεσικής διάταξης που και αυτό είναι ένα ζήτημα εφαρμογής της οδηγίας του 2008 λέει ο πρόεδρος για την οικογενειακή επανένωση, το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Όταν συζητήσαμε και το θέμα των κυρώσεων θα διαπιστώσατε ότι το θέμα ουσιαστικά είναι θέμα κρατών μελών, είναι όμως και θέμα συνθήκης και υπάρχει έτσι, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα με την ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Η οδηγία του 2008 ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, υπό την ήταν σημαντική αυτή η οδηγία. Υπάρχουν όμως προβλήματα υλοποίησης, εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Θα μας πει τώρα τα σχετικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχουν και τι εγκάρσια ζητήματα υπάρχουν, τι προβλήματα εφαρμογής διαπιστώνει για τους νέους συναδέλφους να επαναλάβω ότι ναι μεν είναι θέμα εθνικό κυρίως, εθνικής αρμοδιότητας, αλλά και εμείς επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ευθύνη. Πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση. Να δούμε αντικειμενικά εφαρμόζονται ή όχι σωστά οι οδηγίες αφού ψηφιστούν ή εγκριθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για τη συγκεκριμένη οδηγία θα ακούσουμε την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση αυτής της οδηγίας συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για λόγο ανακοίνωση περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση οδηγία περί δικαιώματο οικογενειακή επανένωση. Και τώρα θυμήθηκα ότι δεν απάντησα κάτι για την οδηγία περί κυρώσεων και αν θα εκδώσουμε κατευθυντήριε γραμμές. Είναι νέα οδηγία από το 2009 πρέπει ε, να έχει εφαρμοστεί στο, στα κράτη-μέλη το 2011. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση, άρα θα ήθελα να σας ζητήσω λίγο χρόνο ε, πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε τον ενδεχόμενο πολύ κυρώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά και τις κατευθυντήριες γραμμές, αυτή οδηγεί ακόμα, ε, μάλλον είναι λιγότερο καινούργια, από το 2003, και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον τομέα αυτό στην Ένωση, γιατί είναι ένα σημαντικό τομέα, αφορά ε, το δικαίωμα οικογενειακή επανένωση ε, για τους μετανάστες και βασίζεται σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα αυτό της οικογενειακής ζωής. Ίσως ε, να είναι αόριστο κάποιες φορές ε, το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής με διάφορες ρήτρε. Δεν υπήρχε και άλλωστε συναπόφαση εκείνη την εποχή. Εγκρίθηκε με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο σίγουρα επηρέασε το περιεχόμενο της οδηγίας. Υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι πολύ αόριστα στη διατύπωσή τους. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της οδηγίας. Να επιτρέψει στα μέλη της οικογένειας υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως να ε, έρθουν να διαμείνουν με τον εν λόγω υπήκο της χώρας. όταν έρχονται ε, υπήκοοι τρίτων χωρών για, σε, για επανένωση και γενική με έναν υπήκο Τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν άλλοι, άλλοι κανονισμοί, άλλες διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας κτλ. Έχουμε κάποια στοιχεία για τα κρατημέλη, τα τελευταία από το 2012, 443.000 επί τρίτων χωρών ε, ήρθαν ε, να επανενωθούν οικογενειακά με υπηκόους τρίτων χωρών για την περίπτωση που ήρθαν ε, για υπήκο της Ένωσης, αυτά τα άτομα ήταν 227.000. οικογενειακή επανένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ο βασικός στόχος της οδηγίας είναι η προστασία της οικογενειακής μονάδας. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που ήρθαν για οικονομικούς λόγους στην Ένωση, πήραν άδεια ε, παραμονής και είναι σημαντικό να έρθει και η οικογένειά τους. Και είναι και σημαντικό να ενταχθούν οι μετανάστες. Με την οικογενειακή επανένωση αυτό ε, διευκολύνει. Και αποφεύγονται άλλες καταστάσεις όπως είναι λευκή γάμη κτλ. Ή πλαστά έγγραφα. Μετά το 2009 είχαμε μια πράσινη βίβλο, έγιναν διαβουλεύσεις, διοργανώθηκε δημόσια ακρόαση με πάνω από 230 ενδιαφερομένους το 2012 και το βασικό θέμα που τέθηκε στην ακρόαση και στη διαβούλευση είναι αν θα πρέπει να αλλάξει η οδηγία περί οικογενικής επανένωσης. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και της ακρόασης. Δεν θα πρέπει να αλλάξει η οδηγία ήταν το αποτέλεσμα. Όμως θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Επτά συναντήσεις είχαμε, έγινε αυτή δηλαδή η ομάδα. Με την κοινωνία των πολιτών ε, και ΜΚΟ, παρότι δεν ήταν ένα αίτημα αυτό, είχαμε επίσης συναντήσεις, γιατί σας φέσω ότι χρειαζόταν και η δική τους άποψη. μελετάμε τους εφιστάμενους ε, κανόνες και τρίτη έκβαση κατευθυντήριες γραμμές που έπρεπε να δημοσιεύσουμε και έχετε και αναχείρα σήμερα. Πρώτα απ' όλα στόχος ήταν να διευκρινίσουμε αυτά τα οποία εντοπίσαμε ως προβληματικά και με τις διαβουλεύσεις. Ο δεύτερος στόχος είναι να υπάρχει διαφάνεια και σαφής κατανόηση των ε, κανόνων και των ε, δικαιωμάτων περικογενικής επανένωσης. Κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών δεν ήταν εύκολη η δουλειά. Είναι πιο εύκολο όταν υπάρχει νομολογία. Δεν ισχύει όμως αυτό στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης, της σχετικής οδηγίας. Τρεις μόνο αποφάσεις ε, δικαστικές έχουμε δύο αποσύρθηκαν και μόνο, μόλις στις 10 Ιουλίου εκδόθηκαν δύο νέες αποφάσεις για την οικογενειακή επανένωση, οι οποίες είναι και πολύ ενδιαφέρουσες. Άρα λίγη νομολογία στην οποία μπορεί κανείς να βασιστεί. Γι' αυτό και εργαστήκαμε με βάση την νομολογία που είχαμε στη διάθεσή μας, εργαστήκαμε με τα κράτη-μέλη και με την κοινωνία των πολιτών για να ολοκληρώσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, Υπάρχουν διάφορες πτυχές, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί νομίζω θα μακρηγορήσω πολύ, αλλά θα περιουστώ σε κάποια σημεία. Διευκρινίζουμε κάποιες πτυχές που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, επί παραδείγματι ο ορισμός ε, ευλόγων προοπτικών μόνιμης διαμονής, ελάχιστη ηλικία συζύγου, διευκρίνηση κανόνων επίσης για την υποβολική εξέταση αιτήσεων, παραδείγματι κατευθυντήριες γραμμές για τα τέλη, συνοδευτικά στοιχεία, πώς αυτά υποβάλλονται, διάρκεια διαδικασίας και τέλος απαιτήσει για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθεαυτού. Ζητήματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, δημόσια υγεία, ε, διαμονή, ασθένεια, ε, υγειονομική περίθαλψη, μέτρα ένταξης, περίοδος αναμονής. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν ε, την είσοδο, διαμονή, διεθνής προστασία, πρόσφυγες κτλ. Είναι αρκετά μακροσκελές και νομικό το κείμενο, αλλά θα έλεγα ότι είναι άρτιο Ακούσαμε τις ε, ΜΚΟ, ακούσαμε την κοινότητα των πολιτών, πήραμε feedback και από τα κράτη-μέλη. Ε, είναι θετικές οι αντιδράσεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημέρωση, πληροφόρηση, ιδίω στα άτομα τα οποία μετοπίζουν δυσκολία στο να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Πολλές φορές υπάρχουν κάποιες προδικαστικές ε, αποφάσεις, ε, διαδικασία υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο κτλ. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή οδηγία με την ομάδα ε, των ειδικών και τη ομάδε επαφή. Έχουμε στείλει επιστολέ προειδοποιητικέ πριν δηλαδή την εκκίνηση μια διαδικασία επί παραβάση. Υπάρχει και μια τέτοια και μελετούμε την νομοθεσία των κρατών μελών Έλαβαμε μία μελέτη την οποία είχαμε αναθέσει για το θέμα αυτό και θα δούμε αν θα χρειαστεί να κινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση. Αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν. Είναι σημαντικό και εδώ το ε, στοιχείο της ενημέρωσης για την οδηγία περικογενικής επανένωσης είναι σημαντική ενημέρωση, όπως και για την προηγούμενη περίπτωση. Πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι μετανάστες να γνωρίζουν επίσης ε, τι δυνατότητες έχουν ώστε να ε, επιβάλλουν το σεβασμό των δικαιωμάτων. Τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμίτς. Ε, μία ομιλήτρια έχουμε, μόνο την κυρία Μπιόρκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ ονόματος της ομάδας μου, Γκουέντζιλ, εμείς θα καλωσορίζαμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Διαπιστώνουμε πάρα πολλές δυσκολίες γιατί έχουμε επαφές με τους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους είναι ανθρώπινο δικαίωμα η πανένωση των οικογενειών, το οποίο τα κράτη-μέλη συστηματικά παραβιάζουν. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή κατευθυντηρίων γραμμών και προσανατολισμών. Βεβαίω, θα θέλαμε να δούμε μια καλύτερη βασική οδηγία με περισσότερα δικαιώματα για την επανένωση των οικογενειών ευθύ εξ αρχή. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώ χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη τι διαδικασίε και τι διοικητικέ διατυπώσεις όταν ζητεί κάποιο να ενωθεί με την οικογένειά του. Τα προβλήματα που υπάρχουν Ε, συχνά προκαλούνται ε, γιατί τους ζητούν οι αρχές διάφορα έγγραφα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν που δεν υπάρχουν καν. Και οι πρεσβείες έχουν τελείως διαφορετικές διαδικασίες κάθε φορά και δεν ξέρουμε ποια είναι και η νομική ασφάλεια που παρέχουν αυτά τα έγγραφα για τους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν τις οικογένειές τους. Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες που πέφτουν θύματα της λεγόμενης έμφυλης βίας και έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα ακόμα και αν εγκαταλείψουν τον άνδρα που τις κακοποιεί. Ακόμα και όταν είχαν έρθει δηλαδή επειδή ήταν σύζυγοι και κακοποιούνται δεν θα πρέπει να απελάβνονται. Τα κράτη-μέλη δεν σέβονται αυτές τις διαδικασίες. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς πώς προτίθεστε, πώς να το πω, να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πραγματικά θα εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Πώς θα εξασφαλίσετε τον έλεγχο και την εποπτεία ότι ε, ναι. πραγματικά αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά. Πάντα από τα κρατημέλη για την επανένωση των οικογενειών. Μία και μόνη, αλλά πολύ καλή, γιατί ανέφερε όλα αυτά τα θέματα και τα θέματα των εγγράφων, που είναι και τεράστιο ζήτημα και των πιστοποιητικών και πολύ ευαίσθητο γιατί υπάρχει μια τεράστια ας πούμε, γραφειοκρατία που καταπιέζει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Παρακαλώ κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω μιλάμε μόνο για κατευθυντήριες γραμμές, για ήπια νομοθεσία ουσιαστικά και βεβαίω για την ε, συμπερίληψη και της υπάρχουσας νομολογίας μπορεί να υπάρξουν και άλλες δικαστικές αποφάσεις, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο εγγύς μέλλον. Και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για να ε, εξετάσουμε την υλοποίηση τη οδηγίας από τα κρατή μέλη. Ε, εξετάζοντας τις εθνικές νομοθεσίες, θα δούμε κι εμείς, εφόσον έχουμε αμφιβολίες, τι λένε οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά. Οι κατευθυντήριες λοιπόν αυτές γραμμές θα είναι η δική μας αφετηρία για να δούμε πώς ακριβώς ε, υλοποιήθηκε η οδηγία στα κρατημέλη. Ε, τι μέτρα έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη και τι γίνεται με τους ε, με συγκεκριμένες υποθέσεις. Υπάρχουν κάποιες ε, δικαστικές υποθέσεις που ακόμη δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί, δεν έχουμε τη δικαστική απόφαση ακόμη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τι αποφάσεις θα λάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τις λάβει σαφώς υπόψη για την προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας επιτρέπουν να δούμε προσεκτικά και σωστά την νομοθεσία των κρατών μελών. Ελπίζουμε ότι τα κρατη έχουν σεβαστεί ε, την ε, οδηγία στην υλοποίηση, τις κατευθύνες γραμμές μάλλον στην υλοποίηση της οδηγίας. Για την ώρα οι αντιδράσεις, οι αποκρίσεις των κρατών μελών ήταν ε, θετικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ιδίω θεωρούμε ότι και με τις κατευθύνες γραμμές θετικά θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη, αλλά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Σμιτ. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τελευταίο σημείο που αφορά την μετανάστευση από το πακέτο αυτό για την μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υλοποίησή της. Θα έχετε ακούσει ακόμα και καινούργια την περίφημη αυτή μπλε κάρτα, ε, μια οδηγία που εγκρίθηκε το 2009, τότε που απλώς ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Η Προθεσμία για την υλοποίηση τότε ήταν ε, ο Ιούνιος του 2011 και η έκθεση υλοποίηση δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για το 2012 και 2013. Το ιστορικό για την πλεκαρτα κάρτα, όπως τα γνωρίζετε συνάδελφοι, ήταν ενός είδους αντιγραφής ή τέλο πάντων μεταφοράς της ε, λογικής της πράσινης κάρτας των ΗΠΑ στην Ευρώπη δηλαδή να υπάρχουν νόμιμοι διάβλοι για την μετανάστευση των υψηλής μόρφωσης εργαζομένων. Οπότε η υλοποίηση αυτού του νομοθετήματος είναι κάτι που αφορά νομίζω πολλούς. Και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας πει τι πληροφορίες διαθέτει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και εδώ να ξεκινήσω με κάποιες γενικές ε, πληροφορίες διότι το θέμα της αναζήτησης ε, δεξιοτήτων είναι κάτι που ε, αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Δεν θέλουμε μόνο τους, τους εργαζομένους με τα υψηλότερα προσόντα, αλλά υπάρχει σοβαρή ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες περιοχές του κόσμου. Θέλουμε λοιπόν όμως, διάβλους για τη μετανάστευση να προσελκύσουμε υψηλών προσόντων ε, μετανάστες, να οθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά μας. Είδαμε τις ελλείψεις που υπάρχουν ήδη και συνεχίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υφίστανται και γι' αυτό το λόγο η οδηγία για την ε, μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εγκρίθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η έκδοση ε, η διευκόλυνση μάλλον της κινητικότητας των εργαζομένων υψηλοπροσόντων και των μελών των οικογενειών τους με καλύτερες ε, συνθήκες υποδοχής, ε, με ένα συγκεκριμένο καθεστώς, υψηλή προστάσια των δικαιωμάτων τους και μεγάλη κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα κάποια στοιχεία. Το 2012 3.640 ε, ε, μπλε κάρτες εγκρίθηκαν και 1.400 για μέλη οικογένειας. Οι περισσότερες μπλε κάρτες ε, δόθηκαν από τη Γερμανία. Εάν διαβάσετε την έκθεση, αυτό είναι εξισημείωτο. Η Γερμανία το 2012 έδωσε 5.484 μπλε κάρτες. Ενώ ακολουθεί η Ισπανία στη δεύτερη θέση με τα 361 μπλε κάρτες. Βλέπετε τη διαφορά. Μετά υπάρχει μεγάλη μείωση με κάποια κάτι μέλη να μην δίνουν καθόλου μπλε κάρτες. Το 2013 έχουμε επίσημα στοιχεία για 15 κράτη-μέλη από τη Eurostat. Ο αριθμός των μπλε καρτών έχει αυξηθεί σε περίπου 12.499 μπλε κάρτες. Πάλι η Γερμανία δίνει τις περισσότερες με 11.580 ενώ ακολουθεί η Γαλλία. Από πού έρχονται τώρα οι εργαζόμενοι των μπλε καρτών, κυρίως από την Ασία αλλά και από την ε, Αμερικανική Ήπειρο, τη Βόρεια και την Νότια Αμερική. Υπάρχει επίσης αύξηση το 2012 ε, με τον εργαζομένο που από την Ινδία, την Κίνα, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία. Ποια είναι τα βασικά ευρήματα της έκθεσης. Το πρώτο σημείο δεν θα σας ευνηδιάσει μετά από αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των μελών στον αριθμό των μπλε καρτών που που εκδόθηκαν. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το μέγεθος αλλά και με τις οικονομικές συνθήκες που γνωρίζουν τα κρατημέλη αυτά. Προφανώς αυτό έχει συνέπειες και στην έκδοση των μπλε καρτών. Εάν η οικονομική κατάσταση είναι δυσχερή και δεν μπορεί κανείς να προσελκύσει εργαζομένους υψηλών προσόντων από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς θα καλέσει και υπηκόους τρίτων χωρών. Και το μέγεθος βεβαίως του κάθε κράτους έχει σχέση με όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την έκδοση μπλε καρτών και σχετικών αδειών. Λόγου χάρη, πώς έχει διαφημιστεί η μπλε κάρτα στα κρατη Δηλαδή, οι εργαζόμενοι μπορούν να πάνε σε ένα προξενείο και να ζητήσουν την μπλε κάρτα. Ε, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μόνο. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρηση. Υπάρχουν επίσης πολλές ρήτρε δυνητικού χαρακτήρα στην οδηγία. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση εφόσον κάποια κρατήφια μέλη θέλουν να την εφαρμόσουν Οπότε προφανώς οι εργαζόμενοι μπορούν να προτιμήσουν ένα, κάτω, ένα από ένα άλλο. Παραδείγματα, τα άρθρα όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν συγκεκριμένε πολιτικές επιλογές για τις ποσοστώσεις, τον αριθμό τους, των εργαζομένων που θα γίνουν αποδεκτοί. Επίσης η περίοδος ισχύω, η διάρκεια ισχύω της μπλε κάρτας, από ένα χρόνο έως μια πενταετία, τετραετία, πενταετία. Οι διαδικαστικές ε, εγγύησεις, πώς εφαρμόζονται τα όρια, όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την ε, έκδοση της μπλε κάρτας. Και βεβαίως μπορεί τα κρατη μέλη, εφόσον διαθέτουν ήδη κάποιο εθνικό πρόγραμμα, να το διατηρήσουν, εν παραλίλω με το πρόγραμμα για την μπλε κάρτα. Κάτι άλλο που εντοπίζει η ανακοίνωση το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα εθνικά προγράμματα για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλών προσόντων πολλές φορές ανταγωνίζονται το πρόγραμμα της μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα είναι τα κράτη-μέλη που έχουν ειδικέ διατάξεις στην νομοθεσία τους ε, για την μετανάστευση γενικότερα, ενώ επτά έχουν ξεχωριστά στοχοθετημένες πολιτικές ε, για την προσέλκυση μεταναστών. Κάποιοι εντοπίζουν τις προτεραιότητά τους σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως τους ερευνητές, τους ε, συνεργαζόμενους μαθητευόμενους και αυτό βεβαίως η συνεργασία των επιλογών αυτών με το, ο συντονισμός μάλλον των επιλογών αυτών με το πρόγραμμα της μπλε κάρτας μπορεί να επηρεάζει την υλοποίηση της οδηγίας την οποία συζητούμε. Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συζητούμε την οδηγία για τους φοιτητέ και ερευνητέ ε, αυτό το διάστημα, οπότε αυτό μπορεί να επηρεάσει τις εθνικές νομοθεσίες και να υπάρξουν αλλαγέ στο προσχές μέλλον. Κάποιοι τομεί επίσης, κάποιοι τομείς, η πληροφορία, η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ε, η μηχανική, είναι τομείς που ε, αφορούν ιδιαίτερως κάποια κράτη-μέλη, στα οποία δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, το 2013, όπως σας είπα, η Γερμανία εξετούσε 10.580 ε, μπλε κάρτες και μόνο 11 με το εθνικό της πρόγραμμα. Σε άλλα κάτι μέλη η κατάσταση είναι τελείως αντίστροφη. Ε, ε, κάποιοι δίνουν πολύ περισσότερε ε, κάρτε εισόδου και δικαίωμα άδειε διαμονή με το εθνικό του πρόγραμμα παρά βάση του προγράμματο τη μπλε κάρτα. Οι διαπραγματεύσει για την μπλε κάρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν ε, δύσκολε γιατί δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουν όλοι ομοφόνο. Αυτό επηρέασε και το περιεχόμενο τη οδηγία προφανώ. Γι' αυτό και προβλέφθηκε η δυνατότητα να συνεχίζουν να υπάρχουν τα εθνικά ε, προγράμματα. Υπήρξαν κάτι μέλη που ήθελαν να υπάρξει, να επιτραπεί ακόμη ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Και νομίζω ακριβώς ο ανταγωνισμός αυτός είναι κάτι που να το δούμε σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου και θα πρέπει έτσι να διαμορφώσουμε και την εικόνα για το μέλλον. Κάποιες δυσκολίες τώρα στη μεταφορά της οδηγίας, χαμηλό επίπεδο συνέπειας, περιορισμένο περιορισμένος βαθμός προστασίας των δικαιωμάτων και περιορισμένη κινητικότητα. Σε κάποιους το πρόγραμμα κινητικότητας προβλέπεται με την μπλε κάρτα φαίνεται πολύ λιγότερο ελκυστικό από αυτό της ενδευρωπαϊκής κινητικότητας ή των ε, μεταφερομένων εργαζομένων. Ε, τα επόμενα βήματα τώρα. Θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τα κατεμέλη στην υλοποίηση της οδηγίας Ήδη συναντηθήκαμε με πολλούς εκπροσώπους των κρατών μελών, με τις ομάδες επαφής, τελευταία φορά μάλιστα τον Ιούνιο, όπου συζητήσαμε δυσκολίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση. Και επίσης θα συνεχίσουμε τη συλλογή πληροφοριών. Πληροφορίες για κάποιες πτυχές που δεν τις καλύπτει τόσο καλά η έκθεση. Δεν είχαμε γέρος όλες τις πληροφορίες λόγω χάρη για τα ε, όρια των αμοιβών, για τους όρους υποδοχής, για την επιστροφή και το κόστος της επανείς για, την, ε, ε, πρόσληψη, για τις διαδικασίες πρόσληψης και το καθεξής. Όπως είπα, οι πληροφορίες εδώ είναι πολύ σημαντικές και εργαζόμαστε σκληρά για τα θέματα μετανάστευση του ή τη τη Ευρωπαϊκή και τα σχετικά προγράμματα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και εδώ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε κύριε Σμιτ. Για το συναδέλφου που δεν ήταν εδώ όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυτή για την μπλε κάρτα, ξεκίνησε πολύ πριν, ε, στην προηγούμενη Ιταλική Προεδρία και υπάρχει εδώ κάποια συμμετρία στην εξέλιξη του θέματος, κάποια αρμονία μάλλον. Όταν ξεκίνησε η, όλη, η όλη συζήτηση για την μπλε κάρτα, θυμάμαι ότι μιλούσαμε για μια ευρωπαϊκή πράσινη κάρτα και πολύ μικρούς αριθμούς τότε. Η Γερμανία ήταν πολύ συνεπή στο σεβασμό των ε, κανόνων, αλλά τελικά οι αριθμοί για τους οποίους συζητούμε είναι τόσο και όντω, όπω είπατε κι εσεί, κάποια από τα εθνικά συστήματα συγκρούονται με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την μπλε κάρτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα μπορούσε να μας πει κιόλα εάν η μπλε κάρτα ενδεχομένως δεν τα πήγε καλά λόγω της λιτότητας γιατί ξεκίνησε πολύ κοντά χρονικά με την έναρξη της κρίσης. Δεν είσαστε πολλοί από σας εδώ όταν ξεκίνησε η όλη συζήτηση. Ε, ήταν κάτι που σκοπό είχε να διευκολύνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κάτι που θα μας οδηγούσε στο να, γίνει, να κάνουμε μια διαλογή ε, από τις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας έλεγε κιόλας εάν υπήρχε μια τέτοια τάση, αλλά τελικά οι αριθμοί είναι αμεληταίοι. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχιστεί και όλα η σχετική προσπάθεια και η έντονη παρακολούθηση του θέματος, διότι τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη η απήχηση του συστήματος αυτού. Η κυρία Κρίσπεκ πρώτη. Ευχαριστώ κυρία και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, συμφωνώ με αυτά που λέτε και με τη διαπίστωση, εν μέρει όμως με το συμπέρασμα μόνο, διότι μπορεί κανείς να φανταστεί ότι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες θα μας είχαν οθήσει να είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι για αυτό το ε, σχήμα που είχαν ζητήσει πολλοί Ευρωπαίοι πριν από 9 χρόνια. Μετά από μια πενταετία εφαρμογής λοιπόν αυτού του συστήματος ε, που ήταν πολλά υποσχόμενο ή περιμέναμε πολλά, ερχόμαστε να το αξιολογήσουμε. Θυμίζω ότι ε, τότε το Κοινοβούλιο είχε μόνο διαβούλευση. Ε, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Χαίρομαι για την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτής της έκθεσης, αλλά οφείλω να πω ότι κάπως έχω απογοητευτεί από τα συμπεράσματα της παρουσίασης. Πέντε χρόνια μετά λοιπόν ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στο σχήμα αυτό. Είπατε κι εσείς Πρόεδρε ότι τα αποτελέσματα ήταν μάλλον αμεληταία και μάλιστα βλέπουμε τεράστια απόκληση. Υπάρχει ένας πίνακας που επισυνάπτεται στην έκθεση και θα εξηγεί πολύ ωραία, τα είπε και η κυρία Σμιτ. Έχουμε τεράστιες αποκλήσεις. Και σε αιτήσια βάση, μάλιστα, για τις κάρτες που χορηγεί και η ίδια χώρα, ας πούμε, στη Γερμανία, ε, από 205 κάρτες ε, γαλαζίες έχουμε περάσει πάνω από 14.000 τον επόμενο χρόνο. Ε, άλλα κράτη-μέλη δεν εκδίδουν ούτε μία μπλε κάρτα το χρόνο. Καμία. Μηδέν. Δηλαδή τα αριθμητικά αυτά στοιχεία είναι πραγματικά έκπληξη προκαλούν σε σχέση με ένα μέτρο ή σύστημα που κανονικά θα έπρεπε πολύ γρήγορα να απογειωθεί. Ε, για τα νομικά ζητήματα το καθεστώς είναι απλό, είναι δεδομένο, οι διαδικασίες απλουστευμένες. Προσπαθήσαμε να εξισορροπήσουμε αυτό για να φρενάρουμε κάπως την ε, ε, φυγή εγκεφάλων και να υπάρχει απαραίτητη άμυλα και ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Το θυμήσατε κι εσείς Πρόεδρε, προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε την Αμερικανική ε, Πράσινη Κάρτα που είναι πραγματικά ένα ε, θαυμάσιο κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη και προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Ε, υπενθύμησε η κυρία Σμίτ ότι οι εθνικές νομοθεσίες είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους αφενός και αφετέρου είναι κακή η εφαρμογή της οδηγίας γιατί έχει μεταφερθεί ε, με λάθος τρόπο στην εθνική νομοθεσία. Αυτά είναι εμπόδια που είμαστε συνηθισμένοι να βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια. Και δεδομένης της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη και πολλών κρατών μελών, ε, και μεταξύ αυτών είναι και δική μου πατρίδα η Γαλλία, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα κάπως να επιταχύνουμε. Και λυπάμαι, ε, καταλήγοντας, λυπάμαι που η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καταλήγει σε αυτό. Ε, παραμένει στις διαπιστώσεις. Ωραία, συμβαίνει αυτό και από εδώ και μπρο τι θα κάνουμε. Α, τι να κάνουμε, δεν λειτουργεί, δεν έχει πιάσει το μέτρο, είναι αλλαντάλλων κατάσταση από χώρα σε χώρα. Μα έχει περάσει μια πενταετία που έχει μεταφερθεί σε όλα τα κράτη-μέλη στην νομοθεσία. Ε, έχει ελλείψει σε αυτό το σύστημα και ζήσαμε και μια προεκλογική εκστρατεία που έγινε μέγας λόγος για ε, το μεταναστευτικό με πολλές συγχύσεις ε, πάντα εις βάρος της Ευρώπης ενώ ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευνοϊκό και ευπρόσδεκτο από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήθελα εγώ να δω και προτείνω στην κυρία Σμιτ χωρίς να ξανανοίξει η οδηγία δεν χρειάζεται θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάμεσα, ε, απέναντι σε αυτή την ανισχυτική κατάσταση, αμεληταία αποτελέσματα που είπατε, να δούμε τι να κάνουμε. Ξέρω και εγώ, να, να προτείνουμε κάτι. Soft law, δεν χρειάζεται να είναι νομοθεσία. Με κάποιες ρυθμίσεις, ας πούμε, κατευθυντήριες γραμμές που κάπως να τονώσουν ε, ε, αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Πολλού δε μάλλον που ο επόμενος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, διατράνωσε σε όλες τις πολιτικές ομάδες τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης για να έχουμε τέτοιους διάβλους και να προσελκύουμε νόμιμους μετανάστες στην Ευρώπη, γιατί τους έχουμε απολύτη ανάγκη. Χαίρομαι για την έκθεση, αλλά έχω απογοητευτεί από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Και θα παρακαλούσα να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτού του συστήματος. Ουσιαστικά. Ή αλλιώς να το καταργήσουμε. Ευχαριστώ, Ναταλή. Ε, θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπαμε και στην αρχή της συζήτησης. Τώρα αρχίζει η συζήτηση. Τώρα θα πρέπει να έχουμε μία αφήγηση για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ε, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να θυμίσω πάλι στους συναδέλφους ότι το βασικό σύστημα ε, από την μπλε κάρτα και που φαίνεται με την έκθεση ε, είναι ότι υπάρχουν εθνικά συστήματα για την είσοδο και την υποδοχή εργαζομένων με συγκεκριμένη ειδίκευση. Ε, Τα εθνικά συστήματα συγκρούονται με τη γαλάζια αυτή κάρτα. Άλλο η πράσινη κάρτα στι ΗΠΑ είναι τελείω διαφορετικό το σύστημα, οι νοοτροπίε, οι μέθοδοι. Δηλαδή το όραμα ή το όνειρο για μια τέτοια μπλε κάρτα ήταν διαφορετικό. Η πραγματικότητα τώρα έρχεται και συγκρούεται με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς αναφέρει μια κατάσταση που ήταν αναπόφευκτο να συμβεί. Τώρα εμείς θα πρέπει να προτείνουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι μοιραίο να το καταργήσουμε γιατί κάποια στιγμή ε, θα μας φέρει σε δύσκολη θέση ή θα το διασώσουμε για να λειτουργήσει σωστά. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα αρχίζει η συζήτηση. Συγγνώμη που προκαλώ λίγο ή προβοκάρω, αλλά γιατί και αλλιώς τα κράτη-μέλη τα δικά τους κάνουν. Η κυρία Σίπελ από τη χώρα που προσπαθεί να κάνει αυτό το σύστημα να λειτουργήσει πάνω κάτω. Τώρα αυτό το τελευταίο ας μην το σχολιάσω. Γιατί ακούγεται θετικά αυτό με τα νούμερα, αλλά μπορεί κανείς να το δει και αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι η διπλή ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Μπλε Κάρτας και των εθνικών διαδικασιών και απαιτήσεων. Υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη τις δικές τους ρυθμίσεις και δεν χρησιμοποιούν αυτή τη γαλάζια κάρτα γιατί τους παρά είναι περίπλοκοι, λιγότερο ελκυστικοί ή γιατί έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις που είναι εξίσου καλές οπότε σου λέει τι να το κάνω, δεν μου χρειάζεται αυτό, είναι περιττό να χρησιμοποιήσω το σύστημα της μπλε κάρτας. Και θα ήταν χρήσιμο να αντιπαραθέσουμε εδώ κάποια αριθμητικά στοιχεία. Όταν λέμε σε πολλές χώρες δεν δίνουν καμία, άλλες χώρες δίνουν πάρα πολλές. Αλλά θα πρέπει να δούμε στις άλλες χώρες πώς συμβαίνουν με τις εθνικές ρυθμίσεις, τις παράλληλες ή ανταγωνιστικές. Και υπάρχουν ε, και συγκρίσεις για το πόσο περίπλοκη είναι η διαδικασία της Βλέ κάρτας σε σύγκριση με τις εθνικές διαδικασίες και ποιες είναι οι υποθέσεις για την υποδοχή ε, ε, υψηλής συνδίκευσης εργαζομένων. Γιατί πολλοί λέγουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική η γαλάζια κάρτα και είναι μάλλον μειονέκτημα στην παγκόσμια αγορά ε, και στον ανταγωνισμό γιατί υπάρχουν άλλες χώρες που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, καλό θα ήταν να συγκρίνουμε αυτή τη γαλάζια κάρτα με τις εθνικές ρυθμίσεις ε, εισόδου στη χώρα και προσέλκυσης εργαζομένων υψηλής συνδίκευσης και να δούμε τι κάνουν και άλλες χώρες εκτός της Ένωσης με τις οποίες βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό. Θα ήταν χρήσιμο και αυτό για να δούμε αν θέλουμε αυτό το σύστημα τη κάρτα να το βελτιώσουμε, αν μπορεί να βελτιωθεί, να το διευρύνουμε, τι θα το κάνουμε, πάση περιπτώσει. Ε, Ευχαριστώ, Μπριγκίτε. Η Τζιν Λάμπερτ την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Έχω κάποια ερωτήματα το πρώτο, με την προσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τρίτες χώρες, σε ποιο βαθμό παρέχουν ενεργά πληροφορίες για το σύστημα της πλεκάρτας. Και δεύτερο, δεύτερο ερώτημα, με τους ίδιους τους ε, οικονομικούς μετανάστες, Υπάρχει κάποια έρευνα ε, που να μας λέει οι ίδιοι τι σύστημα προτιμούν είναι θέμα πολιτικής επιλογής για τα κράτη-μέλη, αν θα προσφέρουν μπλε κάρτα ή ε, σε σχέση με το τα δικαιώματα που έχει το εθνικό σύστημα, αλλά με την μπλε κάρτα υπάρχει και συμπληρωματικά και μια σχετική ελευθερία μετακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα εθνικά συστήματα που πολλές φορές περιορίζουν τον εργαζόμενο σε έναν εργοδότη και σε μια συγκεκριμένη χώρα. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ξέρω, εάν έχετε στοιχεία, για το τι προτιμούν οι ίδιοι οι οικονομικοί μετανάστες, αν βέβαια έχουν την επιλογή. Γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν επιλογή από τα κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει κάποια διαφορά στο... στους ορισμούς. Νομίζω τότε το είχαμε συζητήσει γιατί υπάρχει ε, το θέμα υψηλή δίκευση ή υψηλά προσόντα. Είναι, ίδιο, ε, το, είναι η ίδια διατύπωση και σημαίνει το ίδιο. Κατά ανάγκη όχι μάλλον. Δηλαδή αν θέλουν, αν μάλλον με όπως ορίζεται στην μπλε κάρτα, ε, ο εργοδότης είναι αυτός που αποφελείται γιατί μπορεί να διαλέξει τα προσόντα ε, ή τον εργαζόμενο που επιθυμεί. Σεσίλ Γκέγκε είναι η επόμενη. Ε, Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα δεδομένου ότι και η Ιταλία έχει συμμετάσχει στην έγκριση αυτή τη οδηγία, οπότε και εμείς θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Πιστεύω ότι η μπλε αυτή κάρτα, η γαλάζια κάρτα, δεν έχει λειτουργήσει αρκετά καλά για τους λόγους που αναφέρει και η ε, ανακοίνωση. Υπάρχει και έλλειψη πληροφοριών και αυτό το βλέπει κανείς εάν ρωτήσει τον κόσμο βλέπω ότι δεν είναι γνωστή η μπλε κάρτα. Νομίζω αυτό που τελικά έβλαψε περισσότερο την οδηγία ήταν η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν όπως θέλουν το σύστημα αυτό βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας. Αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα, διότι οι εθνικές νομοθεσίες δεν επιτρέπουν σε όλες τις συνθήκες την ε, υποδοχή ε, υψηλών προσόντων μεταναστών. Όπως είπε προηγουμένως και η συνάδελφος, πρέπει να δούμε τι είδους εργασία θέλουμε να καλύψουμε με την έλευση αυτών των μεταναστών. Ε, κοιτάζοντας τους αριθμούς βλέπουμε ότι δεν αφορούν οι αριθμοί αυτοί μόνο ε, εργαζομένους με υψηλά προσόντα. Μπορεί να είναι κάποιοι που έχουν έναν ε, τίτλο εκπαιδευτικό αλλά χωρίς να είναι κάτι που ανταποκρίνεται ακριβώ τι απαιτήσει των υψηλών προσόντων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να κάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει πώ να βελτιώσει το σχετικό σύστημα και όχι να το εξαλείψει. Ακόμη και σε περίοδο κρίση ε, θα πρέπει να μπορούμε να καλύψουμε καταπηγούσε ανάγκε. Δίνω το παράδειγμα τη Ιταλία, όπου εμεί πρέπει να εργαστούμε κάπως ε, πιεσμένα και σε αυτήν την περίοδο να καλέσουμε στην επικράτειά μας και εργαζομένους ε, υψηλής μόρφωσης, με υψηλά προσόντα, οπότε να αλλάξουμε και κάποιους ε, εθνικούς μας κανόνες. Το να δούμε τι μπορεί να γίνει με την πρόληψη, τι μπορεί να γίνει με το θέμα του φαινομένου της μετανάστευσης γενικότερα, είναι κάτι που η γαλέζια κάρτα μπορεί να μας διευκολύνει να το κάνουμε, διότι μπορούμε να φέρουμε περισσότερους εργαζομένους με νόμιμους διάβλους στην επικρατειά μας. Μιλάμε για εργαζομένους μετανάστες που έρχονται στην επικράτεια να έρθουν ε, στην ε, χώρα και να υποβληθούν στην εθνική νομοθεσία. Αλλά με άδειες πραμονής που είναι αιτήσει και πρέπει να ανανεώνονται κάθε χρόνο. Κάποιοι έρχονται λίγο καθυστερημένα λόγω του συστήματος και αυτό βεβαίως αποθαρρύνει τους ε, εργαζομένους με ψηλά προσόντα που Μπορεί να θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, αλλά θα το σκεφτούν. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε εδώ σε τρία σημεία. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα αυτό μόνο σε κατεπίγουσε συνθήκε. Ε, το σύστημα τη μπλε κάρτα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάζουμε τα κριτήρια κάθε φορά, αλλά θα πρέπει μόνιμα ε, να κοιτάξουμε να αποφεύγουμε ε, επεισόδια όπως τα πρόσφατα που είδαμε στην Ιταλία ή το παράδειγμα της Γερμανίας σε περίοδο κρίσης, βλέπουμε ότι δεν δείχνει σχετισμό τη ανεργίας με το χρήση του συστήματο τη γαλάζια κάρτα. Βλέπουμε ότι ο λαϊκισμό αναφέρεται στου μετανάστε και του διασυνδέει με την ανεργία. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι οι άνεργοι δεν είναι ε, όσοι θα είχαν την ίδια δουλειά αλλά μπορεί να απασχολούνται σε διαφορετικούς τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε και τη δική μας την προσέγγιση, την δική μας τη φιλοσοφία. Εγώ θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί την εφαρμογή του συστήματος και σε άλλες χώρες να μην αφήνει τέτοια, να μην προβλέπεται το σύστημα με προαιρετικούς όρους, αλλά να φέρουμε στην Ευρώπη την, ε, ακριβώς την ε, μετανάστευση και τους εργαζομένους που χρειαζόμαστε. Το σύστημα της μπλε κάρτας θα πρέπει να μας φέρει επίσης και στο θέμα της διεθνούς συνεργασίας. Εάν δούμε τα δεδομένα θα καταλάβουμε ότι οι περισσότερες μπλε κάρτες ε, που αφορούν εργαζομένους αφορούν μάλλον εργαζομένους που έρχονται από χώρες από περιοχές της Ασίας ή της Αφρικής. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην πηγή λοιπόν στις χώρες αυτές. Η γαλάζια κάρτα μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε το θέμα αυτό, να στηρίξουμε ενδεχομένω και άλλε πολιτικέ με ευρύτερο προσανατολισμό όπω τη διεθνού συνεργασία, ε, την εξωτερική μα πολιτική. Γιατί από την Αφρική είναι ελάχιστοι εργαζόμενοι που έρχονται εδώ και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι που απασχολούνται ε, παράνομα και μπορεί να έχουν ένα δίπλωμα, μπορεί να έχουν κάποιο πτυχίο, αλλά δεν διαθέτουν τη γαλάζια κάρτα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο όλο σύστημα μια προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Σεσίλη. Στην έκθεση ε, δεν υπάρχουν πολλά που να συνδέουν ακριβώς τις χώρες ε, καταγωγής ή αποστολής με αυτή τη διαδικασία της μπλε κάρτας και χρειαζόμαστε πιο πολλές λεπτομέρειες σίγουρα. Η Άννα Γκόμες είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι δεν αμφιβάλλω καθόλου για το ότι ένας από τους λόγους τους οποίους δεν χρησιμοποιείται περισσότερο η μπλε κάρτα είναι γιατί υπάρχει πράγματι κρίση στην Ευρώπη. Ότι δηλαδή πολλές χώρες δεν χρειάζεται να, να ζητήσουν αλλού ε, Υψηλή ειδίκευση, εργατικό δυναμικό, γιατί έχουν ε, φυγεί εγκεφάλων από τη δική τους χώρα. Όπως στην Πορτογαλία τη χώρα μου, εμείς εξάγουμε ε, τους ικανότερους δημόσιους υπαλλήλους και άλλους επαγγελματίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ιδίω στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη για, τις, ε, για τους γιατρούς. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Νορβηγία συχνά έρχεται εδώ για να, στη χώρα μου, δηλαδή την Πορτογαλία, για να προσλάβει υψηλή ειδίκευση επαγγελματίε. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι και άκρο αρνητικό και κακό, γιατί έχει τεράστιε επιπτώσεις για την ανάπτυξη της χώρας μας. Η μπλε κάρτα είχε ως στόχο αρχικά ε, να προσελκύει εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ε, διαστρεβλώνεται ε, το αποτέλεσμα. Πώς βλέπει η Κομισιόν τη σχέση με αυτή την τεράστια οικονομική ύφεση και αυτές τις μεγάλες ε, ανισότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε το πρόβλημα αυτό και σε ποιο βαθμό το υφιστάμενο σύστημα, μπλε κάρτα, πώς να το πω, διευκολύνει τη νομιμοποίηση των, τρίτων, των επικών τρίτων χωρών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υψηλή δίκευση και θα μπορούσαν πράγματι αν αναγνωριστούν ε, οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους να χρησιμοποιηθούν. να είναι υποψήφιοι για την μπλε κάρτα, αναφέρομαι στη χώρα μου την Πορτογαλία, που είχαμε και έχουμε πολλούς αλλοδαπού από την Ουκρανία για παράδειγμα και άλλες χώρες άτομα με υψηλή δίκευση που εργάζονται όμως ε, σε όχι τόσο σημαντικές θέσεις εργασίας γιατί δεν έχουν αναγνωριστεί οι ικανότητες και τα προσόντα τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για άλλους λόγους ε, ως ε, πρόσφυγες και Δεν θα έπρεπε να γνωριστούν τα προσόντα αυτών μέσω και της διαδικασίας της μπλε κάρτας. βέβαια αυτό που με ανησυχεί πολύ περισσότερο από την μπλε κάρτα, και όχι δεν μιλάω μόνο για την Πορτογαλία, είναι κάτι που ε, λέγεται χρυσή βίζα, η χρυσή θεώρηση που χορηγείται. Αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θετικό αυτό που συμβαίνει τελευταία. Θα ήθελα να το ερευνήσει λίγο η Κομισιόν για να δει τι τεράστιες ε, συνέπειες έχει αυτή η διαδικασία, γιατί με τη Χρυσή Βίζα εισάγουμε εγκληματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Το 2011 ετέθησε σε ισχύ αυτή. Ε, είναι δύσκολο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πώς θα ήταν η κατάσταση εκτός λιτότητος ε, σε άλλη οικονομική συγκυρία. Γιατί άρχισε να εφαρμόζεται με σούσεις της λιτότητος. Η κυρία Σεμπάγιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία καλύπτει μόνο ε, τους εργαζόμενους ε, η, υψηλή δίκευση. Όπως σας είπα προηγουμένως, είχαμε διαφορετικό σύστημα στη Σουηδία το 2008 ε, ε, άρχισε να εφαρμόζεται ένας νόμος για την μετανάστευση και την απασχόληση που κάλυπτε και ανειδίκευτους και ε, ειδικευμένους και μάλιστα υψηλή ειδίκευση εργαζομένους και μετανάστες. Πρέπει να σας πω ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση και ίσως είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Σουηδία έχει εκδώσει τόσες λίγες γαλάζιες κάρτες μέχρι σήμερα. Αν ε, συνυπολογίσετε όμως ε, το σύνολο, είμαστε σε καλή θέση και στον πίνακα 3 που συγκρίνει τις διάφορες εθνικές ρυθμίσεις θα διαπιστώσετε ότι και μάλιστα ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε νομοθεσία που να καλύπτει όλους τους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη για να βρουν δουλειά, χαμηλής και υψηλής ειδίκευσης. Στο μέλλον χρειαζόμαστε νομοθεσία που να μην καλύπτει μόνο τους σούπερ ειδικού ή τους εμπειρογνώμονες, αλλά όλους τους εργαζόμενους που μεταναστεύουν για να εργαστούν στην Ευρώπη. Όταν εισήχθη το σύστημα της γαλάζιας κάρτας, θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ εγωιστικός τρόπος αυτός να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση το εργατικό δυναμικό που χρειαζόταν. Ε, και να διαλέγει ε, τους ε, πλέον ειδικευμένους, τους καλύτερους, ενώ ήθελε τόσο κόσμος να έρθει να εργαστεί. Από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου συχνά. Ε, Εμεί θέλουμε βοήθεια, αλλά οι ανάγκε είναι πολύ μεγαλύτερε. Χρειαζόμαστε μια ανοιχτή αγορά εργασία, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λόπε Αγγιλάρ. Χουάν. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Κομισιόν, η οποία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η συνάδελφός μας μόλις τώρα, η Άννα Γκόμες. Θα γνωρίζετε ότι αυτή την αρνητική στάση προς την νόμιμη μετανάστευση την παρακολουθούμε εδώ και χρόνια και κυρίως αυτά τα χρόνια που ισχύει αυτή η οδηγία από το 2009 και μετά, οπότε δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μέσα από τη χειρότερη κρίση που έχει βιώσει ποτέ στην ιστορία της. Το σημείο λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι σε ό,τι αφορά την έλλειψη αποτελεσματικότητας αυτής της οδηγίας έχουμε να διδαχθούμε πολλά. Πρώτα απ' όλα ότι τελικά στόχο είχε ε, τη φυγή εγκεφάλων άτομα υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες. ενώ απ' την άλλη έχουμε την οικονομική εξορία ανθρώπων ε, επίσης με πολύ ψηλά προσόντα, από φύτους πανεπιστημίων, τεχνικών σχολών, ε, ιδίως από τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να Γκόμες μίλησε για την Πορτογαλία, εγώ μπορώ να σας μιλήσω για την Ισπανία. Αυτή την οικονομική εξορία τη βλέπουμε. Κατοντάδες χιλιάδες ε, νέοι με πάρα πολλά προσόντα πολλοί από αυτούς ξενιτεύονται. Θέλω λοιπόν να, να ρωτήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ανέφερε αυτά τα νούμερα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι καταφέρνουν ε, στη χρήση του συστήματος της μπλε κάρτας. σε σχέση με τον αριθμό και τα προσώτα των ατόμων που μεταναστεύουν σε μια άλλη χώρα μέλος της Ένωσης. Για να καταλάβουμε καλύτερα την αναλογία. Και μήπως αλλάξει και η διάθεση ε, σε σχέση με την έγκριση του πακέτου για την μετανάστευση που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Γιούγκερ εντός επόμενης πενταετίας. Ευχαριστούμε. Ε, πρέπει να δούμε και τι μορφή θα πάρει η νόμιμη μετανάστευση ή η λάθρο μετανάστευση με τα νέα μέτρα. Η κυρία Βεζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά είναι αυτά που ήδη υπόθηκαν και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι κάποιες διαπιστώσεις είναι αναπόφευκτες. Αλλά κάτι στο οποίο μπορεί να μην συμφωνήσουμε είναι ότι μας απογοητεύουν τα συμπεράσματα. Τίνω να πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο να είναι απογοητευτικά. Εδώ και κάμποσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά βρίσκει διαφορετικά συστήματα και τα πολλαπλασιάζει και τελικά τις ευθύνες τις διατηρούν τα κράτη-μέλη. Από το παράδειγμα της Γερμανίας κατάλαβα ότι η ενισχύθηκε το σύστημα της μπλε κάρτας, τα πήγε καλά, αλλά εις βάρος του εθνικού συστήματος ε, υποδοχής μεταναστών στην Γερμανία. Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικά αυτά τα αποτελέσματα ή μη αναμενόμενα. Για να είμαστε επικοδομητικοί εγώ προσωπικώς ε, πραγματικά με εν μέρη, αλλά όχι και τόσο για τις χώρες προέλευσης. Θα μπορούσαμε αυτή την ανάλυση να την δούμε εκ παραλίλου, διότι σε κάποια κράτη, ιδίως τα κράτη της γειτονίας ε, του νότου της Μεσογείου, με συμφωνίες κινητικότητας, ε, κάνουμε να απηχούν ε, οι δικές μας οι ανάγκες με συμφωνίες κινητικότητας ή συμφωνίες επανεισδοχής που αντισταθμίζουν οι μεν τις συνέπειες των δε. Οι συμφωνίες κινητικότητας παραμένουν ακόμη θεωρητικές. Βλέπουμε τι κριτήρια επιβάλλονται. Είναι ακριβώς τα κριτήρια της, ε, του συστήματος της μπλε κάρτας. Θα έπρεπε λοιπόν να προσπαθήσουμε με κάποια από αυτά τα κράτη να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Γνωρίζω πολύ καλά τα ζητήματα της Τινησίας πολύ συγκεκριμένα και έχω πολλούς συνομιλητές από εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργοδοτών εκεί, με κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στα θέματα αυτά. Θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια συνεπή προσέγγιση στα θέματα αυτά. Ε, με τους ε, πετυτραμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί που γνωρίζουν πολλά γιατί κάποιο άλλο στοιχείο που πραγματικά με ε, είναι αυτό που αναφέρθηκε για την αποστράγγιση, την ε, φυγή των εγκεφάλων όπως λέγονται, των εργαζομένων υψηλών προσόντων προς τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Αυστραλία, την, τον Καναδά. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες χώρες προέλευσης τις δικές μας, διότι έχουν κλείσει οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς. Δεν έχουν πια φοιτητικέ ε, θεωρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άδεια παραμονής, οπότε πάνε αλλού. Θα πρέπει λοιπόν η μελέτη αυτή να γίνει και να δούμε τι νομικό σύστημα θέλουμε να προβλέψουμε. Εγώ δεν έχω αυταπάτες, αλλά έχουμε μπροστά μας κάμποση δουλειά για τα θέματα αυτά ακόμη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λόριστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στομικά. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κυρία Ναγκόμες ε, επέκτηνε ε, τη συζήτηση στις χώρες εκείνες οι οποίες ε, είναι σε πιο δινή οικονομική κατάσταση, με χαμηλούς μισθούς, κάτι που αναγκάζει άτομα με ψηλά προσόντα να εγκαταλείπουν τη χώρα τους και να πηγαίνουν σε άτομα με πιο εύρωστη οικονομία, ε, σε χώρες μέλη της ε, Ένωσης με πιο εύρωστη οικονομία. Αυτό το σύστημα της μπλε κάρτας θα πρέπει να τροποποιηθεί για να είναι δυνατόν τα άτομα αυτά που έχουν μπλε κάρτα να πηγαίνουν στις χώρες με μεγάλη φυγή εγκεφάλου Διότι και στην Εστονία έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Έχουν φύγει πολλοί ε, που έχουν καταλήψει για άλλες σκανδιναβικές χώρες Παραδείγματο χάρη, διαθέσαμε 400 εκατομμύρια για να εκπαιδεύσουμε άτομα με υψηλά προσόντα, τα οποία όμω εργάζονται τώρα σε άλλε σκανδιναβικέ χώρε, παίρνοντα βέβαια τα τριπλάσια χρήματα από αυτά που θα έπαιρναν στη χώρα μα. Και ισχύει αυτό για πολλά επαγγέλματα, γιατρού ε, κτλ. Εγώ λοιπόν ε, θα έλεγα ότι χρειάζεται να προωθήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών που το έχουν ανάγκη. Και όχι να φέρνουμε υπηκός τρίτων χωρών με υψηλά προσόντα. Επίσης, καλό θα ήταν να εκπονήσουμε τα δικά μας εθνικά προγράμματα, που ναι, έχουμε τέτοια προγράμματα, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε με υπερβολικά υψηλούς μισθούς, τουλάχιστον σε σχέση με αυτούς που δίνουν οι Γερμανοί ή Βρετανοί, αυτά τα άτομα με υψηλά προσόντα. Ευχαριστώ. Και εδώ τελειώνει ο κατάλογος των μιλητών και ξαναδούμε το λόγο στην κυρία Σμιτ, αν θέλει να απαντήσει σε ορισμένες από τις ειδικέ ερωτήσεις που έγιναν και είναι και δύσκολο καμιά φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά τώρα για αλλαγή. Για ποιο λόγο η οδηγία δεν είχε τα επιθυμητά και αναμενόμενα αποτελέσματα ή τον αντίκτυπο. Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Κάναμε μια ανάλυση με βάση κάποιους οικονομικούς δείκτες, ε, συγκρίναμε τον αριθμό των μπλε καρτών που χορηγήθηκαν, αλλά αυτό δεν βοήθησε πάρα πολύ στην ανάλυση μας. Ε, είδαμε και άλλους δείκτες, την ανεργία κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα, πολύ δε περισσότερο που και τα στοιχεία που μας δόθηκαν είναι αρκετά σαφή και πρέπει να το πω και αυτό. Επίσης κοιτάξαμε ποια είναι τα κράτη-μέλη που έχουν ε, ποσοστώσεις για την υποδοχή οικονομικών μεταναστών και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί και οι ποσοστώσεις ορίζονται βάσει ε, των αναγκών κάθε χώρας και της κατάστασης της απασχόλησης, της ανεργίας στην εκάστοτε χώρα. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Υπάρχουν μερικά στοιχεία τα οποία ανέφερα και στην προηγούμενη μου τοποθέτηση. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν εθνικά συστήματα πιο ελκυστικά. Ε, έχετε όμως συνημένει στην έκθεση ένα πίνακα που κάνει συγκρίσεις πόσες μπλε κάρτες δόθηκαν και πόσες ε, εθνικές αντίστοιχες κάρτες στις χώρες που έχουν τέτοιο σύστημα. Δυστυχώς σήμερα εγώ δεν μπορώ να σας δώσω μια τελική απάντηση. Θα συνεχίσουμε να αναλύουμε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει γίνει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης για τη μεταναστευτική πολιτική των κρατών μελών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση μεταναστών με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. Το 2013 βγήκε αυτή η μελέτη, θα βρείτε εκεί κάποιες ε, απαντήσεις ίσως όχι όλες. Τώρα, σε ποιους τομείς εργάζονται οι κάτοχοι μπλε κάρτας και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί όταν είναι τόσο χαμηλά τα νούμερα ε, και επίσης και τα κράτη-μέλη δεν σας δίνουν τις στατιστικές, είναι πολύ δύσκολο να καταλήξεις κάπου. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα έχουμε κάποια στοιχεία, μια στιγμή για να τα βρω γιατί τα άχασα τώρα. Νομίζω 133 ήρθαν ε, ως μηχανικοί και επιστήμονες και 76 ε, μάνατζερ. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα ως νούμερο, γιατί δεν έχουμε αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία. Μπορεί η έκθεση να είναι κάπως ε, απογοητευτική, γιατί κάνει διαπιστώσεις και ορισμένους προβληματισμούς εκφράζει που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Ήδη έχουμε αρχίσει, ε, σας είπα, να κοιτούμε πώς θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, τι αντίκτυπο έχει και τι αποτελέσματα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολη η ανάλυση της κατάστασης. Όπως είπε και η κυρία Γκρισμπέκ, ο επόμενος πρόεδρος ε, της Επιτροπής Γιούνκερ ε, τόνισε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ελκυστική. Και ανέφερε και ο ίδιος, ε, ακριβώς επειδή δεν εφαρμόζεται καλά αυτό το σύστημα της μπλε κάρτας, ε, ανέφερε και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας. Ξέρετε, αναθεώρηση μιας οδηγίας δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι ε, κάτι που διαρκεί. Λοιπόν, να δούμε ποιες είναι οι δυναμίες, τι λειτουργεί, να καταλάβουμε γιατί ορισμένες χώρες εκδίδουν περισσότερες μπλε κάρτες, ε, έχει να κάνει με το μέγεθος της χώρας, με την οικονομική της κατάσταση, για να μπορέσουμε καλύτερα να αναλύσουμε την ε, κατάσταση. Και ε, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή για να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ και όπως είπε και ο κύριος Thank ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό που δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και είναι πολύ σημαντικό να μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή και λεπτομερή εικόνα για τα κράτη-μέλη εδώ στην Επιτροπή μας. Είναι πραγματικά κάτι που είναι πολύ απογοητευτικό όταν δεν λαμβάνουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Όμως ευχαριστώ πολύ την κυρία Σμίτ για αυτό το μαραθώνιο παρουσιάσεων για τους τρεις αυτούς τομείς, για τα τρία αυτά νομοθετήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ συνάδελφε για την πολύ πλούσια αυτή συζήτηση. Όπως είπα, ευθύς εξ αρχής θα υπάρξουν εξελίξεις και στους τρεις τομείς ανάλογα με το τι θα γίνει και από την πλευρά των Κοινοβουλίου ως πρόταση. Τώρα, το επόμενο σημείο. Παρουσίαση από την Επιτροπή, αυτή τη φορά από τον κύριο Νίλσελ, μια παρουσίαση εξαμηνιαία που αφορά το χώρο του Σέγγεν και γίνεται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε τώρα την πιο πρόσφατη έκθεση για το διάστημα 1 Νοεμβρίου 2013-30 Απριλίου 2014 και οι συνάδελφοι θα αντιληφθούν ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια η λειτουργία του Σέγγεν, του χώρου Σέγγεν ήταν κρίσιμη σημασία για αυτή την Επιτροπή. Η ρήτρα ασφάλειας του Σέγγεν και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε είχε πολύ μεγάλες συνέπειες και επηρέασε πάρα πολύ τη λήψη αποφάσεων εδώ. Μας απασχολούν διαρκώς λοιπόν τα ζητήματα αυτά. Βεβαίω ε, φαίνονται κάπως τετριμένα αυτά τα καθημερινά ζητήματα, όμως έχουν γίνει ένα θέμα κρίσιμο για τη λειτουργία τη δική μας στην Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρώτη της ε, αυτή εξαμηνία παρουσίαση για φέτος. Κύριε Νίλξε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μα καλέσετε λοιπόν να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση που πολύ σωστά είπατε ότι προσπαθούμε να την καταρτίζουμε δύο φορές το χρόνο για να κάνουμε έναν απολογισμό ε, του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος του Σέγγεν, ε, ένα είδος ε, check-up του Σέγγεν όπως το αποκαλούμε, να εντοπίσουμε προβλήματα, ενδεχόμενες εντάσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων ή μεταξύ κρατών μελών, να έχουμε δηλαδή μια τακτική προγραμματισμένη δυνατότητα να εντοπίζουμε προβλήματα και να προτείνουμε κοινέ λύσεις όπως Ξέρετε, είναι η πέμπτη έκθεση. Το Συμβούλιο πάντοτε προγραμμάτιζε σε επίπεδο υπουργών ε, τη συζήτηση για κάθε έκθεση. Πρέπει να σα πω βέβαια ότι για το Κοινοβούλιο δεν ίσχυε πάντα το ίδιο. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να σα παρουσιάσω αυτή την έκθεση, γιατί απευθύνεται εξίσου και στα δύο όργανα, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Συνολικά και συνοπτικά, τι προσπαθούμε να καλύψουμε με την έκθεση. Τρία πράγματα κυρίω. Πρώτον, να δώσουμε τη γενική εικόνα της κατάστασης στα εξωτερικά μας σύνορα, χρησιμοποιώντας ως το δυνατόν πιο επικαιροποιημένα στοιχεία για την περίοδο που καλύπτει η έκθεση. Δεύτερον, να δώσουμε πληροφορίες για την ε, εφαρμογή του κεκτημένου από τα κράτη-μέλη, ιδίω ε, το κεκτημένο που αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Τρίτον, επισκόπηση ζητημάτων ε, που σχετίζονται με το κεκτήμα του Σέγγεν όπως πολιτική ε, είτε χάραξη είτε εφαρμογή της πολιτικής, ε, το ΣΥΣ2, σύστημα ενημέρωσης, πολιτικές επιστροφών. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία λοιπόν για αυτή την πέμπτη έκθεση, ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα και την κατάσταση δηλαδή πιέσεις, οι παράνομες διελεύσεις. Σας παραπέμπω και στη χθεσινή συζήτηση που είχατε για τη συνέχεια στην ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι οι βασικές μεταναστευτικές πιέσεις εντοπίζονται στην κεντρική Μεσόγειο, διαθαλάσσεις μέσω, μέσα προς την ε, Ιταλία και τη Μάλτα, ή μέσω των διαφορών. Δεν θα επανέλθω για άλλα βήματα των εξωτερικών σύνορων. Θα έλεγα ότι σε σχέση και σύγκριση τόσο με τη Μεσόγειο όσο και με τα προηγούμενα έτη, βλέπουμε να είναι σταθεροποιημένη η κατάσταση, να έχουμε χαμηλά σχετικά επίπεδα ε, πίεσης. Η πίεση μειώνεται, ιδίως ότι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Προσπαθούμε επίσης να σκιαγραφίσουμε λίγο την κατάσταση και εντός του χώρου Σέγγεν. Αποτελεί αυτό πρόκληση βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι πλέον στα εσωτερικά σύνορα. Συνεργαζόμαστε εδώ και κάποιο καιρό με τη Frontex για να Έχουμε στοιχεία της λεγόμενης δευτερογενής μετακινήσεις, δηλαδή υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στο χώρο Σέγγεν, πώς μετακινούνται μεταξύ των χωρών. Ε, κάναμε κάποια πρόοδο στον τομέα αυτό, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια από τα κρατη δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από τα κράτη-μέλη, ώστε η Frontex να αναλύσει την κατάσταση καλύτερα και να μας δώσει και εμάς ε, την εικόνα αυτών των δευτερογενών ε, μετακινήσεων εντός του χώρου Σέγγεν. Αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε καλύτερα την όλη λειτουργία του χώρου Σέγγεν των ενδεχόμενων επιλογών ε, κράτων μέλων. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κεκτημένου και ξεκινώ με τα αστερικά σύνορα. Στη διάρκεια της περίοδου αναφοράς είχαμε δύο υποθέσεις όπου προσωρινά επανεισήγαγαν ε, ελέγχους στα αστερικά σύνορα τα κρατημέλη, ε, η Πολωνία για δύο εβδομάδες σε σχέση με μια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και η δεύτερη χώρα ήταν η Ολλανδία, πάλι για δύο εβδομάδες σε σχέση με τη διάσκεψη κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια. Και εκτός της περίοδου αναφοράς είχαμε πανεισαγωγή από το Βέλγιο για έξι ημέρες, αρχές Ιουνίου, των ελέγχων, επειδή υπήρχε η διάσκεψη κορυφής της ομάδας των 7 κοινοποιήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις αυτές οι επανεισαγωγές των ελέγχων ε, στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη και στην περίπτωση της Πολωνίας τουλάχιστον ε, είχαμε και αναφορά για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Γενικά λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει κάποια ένσταση ή αμφισβήτηση. Σε ό,τι αφορά την διερεύνηση πιθανών καταγγελιών ή παραβάσεων από τα κράτη-μέλη, στις εκθέσεις αυτές ε, συνήθως καλύπτουμε ε, πρώτα απ' όλα ε, αστυνομικούς ελέγχους σε ζώνες εσωτερικών συνόρων. Είναι έλεγχοι οι οποίοι επιτρέπονται, όπως γνωρίζετε, αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο των συνοριακών ή τελωνιακών ελέγχων, Είχαμε κάποια παράπονα ή καταγγελίες πολιτών οι οποίοι όταν, όταν ταξίδευαν υποβλήθηκαν σε τέτοιους ελέγχους. Διερευνούμε επίσης πιθανά εμπόδια στα εσωτερικά σύνορα. Για παράδειγμα, ε, όταν ε, ένας αυτοκινητόδρομος διασχίζει εσωτερικά σύνορα μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιες, κάποια ώρα κυκλοφορίας ή κάποιες πινακίδες. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο βρίσκονται, αν είναι θέμα υποδομής, αλλά όχι γιατί περνάει αυτός ο αυτοκινητόδρομος από εσωτερικά ε, Επίσης εξετάζουμε και τη διαδικασία, τις διαδικασίες επί παραβάση ή προκαταρκτικές διαδικασίες, αν υπάρχουν. Έχουμε μια υπόθεση ανοιχτή ε, σε ό,τι αφορά εδώ ε, Σέγγεν πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξει η νομοθεσία για την ευθύνη των αερομεταφορέων, γιατί αυτό πρέπει να ισχύει μόνο για τα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε ζητήσει από το κράτο μέλο λοιπόν να προβεί σε αυτή την αλλαγή. Επίση, έχουμε τρει υποθέσει με τα κρατημέλη για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εξωτερικά σύνορα. Και σε μία περίπτωση ένα κράτος μέλος ελεύθερη διακίνηση προσώπων και ώρα αναμονής, χρόνος αναμονής για τη διέλευση των συνόρων. Αυτά είναι ανοιχτά. Άλλα θέματα που μπορούμε να αναφέρουμε για την κατάσταση. Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την απόφαση περί άρσης ε, ε, των ε, ελέγχων με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό γιατί έχουν περάσει τα κριτήρια και τις αξιολογήσεις σε αυτά τα δύο κράτη-μέλη, αλλά βέβαια εναπόκειται στο Συμβούλιο να πάρει τη σχετική απόφαση. Ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι ότι και εσωτερικά σε επίπεδο Επιτροπή, αλλά και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ξεκινήσαμε την υλοποίηση ε, του τρίτου μηχανισμού αξιολόγησης έγκεν που συμφωνήσαμε τον, το φθινόπορο του 2013. Τέθηκε σε ισχύ ο νέος μηχανισμός αλλά από τις 27 Νοεμβρίου του τρέχοντος θα αρχίσει η πρακτική του εφαρμογή. Μέχρι στιγμής έχουμε γκρίνει το πολιετές πρόγραμμα, το οποίο καθορίσει το χρονοδιάγραμμα, ποιο κράτος μέλος θα αξιολογηθεί και πότε ε, στη διάρκεια της περίοδου 2015-2019 και επίσης και το πρότυπο ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις αξιολογήσεις ε, και για όλους τους τομείς και του κοινοτικού, μάλλον του κεκτημένου Σέγγιν το έχουμε οριστικοποιήσει. Επόμενο βήμα θα είναι η έγκριση του ετήσιου προγράμματος για το 2015 όπου θα αναφέρουμε ε, πιο αναλυτικά τα αξιολόγηση, μάλλον το πρόγραμμα αξιολόγηση των πέντε κρατών μελών για αυτό το χρόνο και τις, ε, μη, μάλλον αυτές τις ευνηδιαστικές επισκέψεις που θα κάνουμε σε οποιοδήποτε άλλο κρατοσμένος και όχι μόνο στα πέντε αυτά. Έχουμε ζητήσει επίσης ε, και input από τη Europol, από τον Οργανισμό Θεμελιτών Δικαιωμάτων ε, και τη Frontex για να εντάξουμε τα σχετικά στο τέτοιο μας πρόγραμμα το Νοέμβριο φέτος. Για άλλα, άλλα θέματα της έκθεσης. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Κάνουμε μια επισκόπηση της λειτουργίας του συστήματος ε, πληροφόρηση και της θεωρήση στη δεύτερη γενιά του ΣΥΣ, συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Για το ΒΙΣ έχουμε ένα επικαιροποιημένο στοιχείο από 1η Απριλίου. 6,7 εκατομμύρια αιτήσει θεωρήσεων έχει επεξεργαστεί το σύστημα. Ε, φτάνουμε στο τέλος μιας νέας μεταβατικής περίοδου, το φθινόπωρο, που τα κράτη-μέλη συστηματικά θα πρέπει να ελέγχουν ε, τα αποτυπώματα στο ΒΙΣ όταν ε, υπάρχει διέλευση εξωτερικών συνόρων. Από τον Οκτώβριο του 2014 το έχουμε πενθυμίσει στα κράτη-μέλη αυτό το νέο καθήκον. Επίσης κάναμε έναν απολογισμό της διευκόλυνσης ή απελευθέρωσης θεωρήσεων. Σημειώνουμε ότι η κατάσταση με άτομα τα οποία έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια και αιτούνται άσυλο, η κατασταση με ατομα που ερχονται απο προβληματική και τουνται ασυλο η κατασταση παραμενει προβληματικη και εξακολουθουμε να την παρακολουθούμε. Δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες ε, για τα υπόλοιπα σημεία της έκθεσης, αλλά αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, να σας πω πρώτα απ' όλο ότι η έκτη έκθεση είναι προγραμματισμένη όπως πάντα για τον Νοέμβριο. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Νίλσεν. Να πω για τα νέα μέλη ότι αυτό το check-up του Σέγγεν γίνεται δύο φορές το χρόνο. Αλλά αυτή η προσωρινή επανεισαγωγή ελέγχων ειστερικά σαν ήταν ένα πραγματικό τεστ, μια πραγματική δοκιμασία για την Επιτροπή μας ε, και γενικώ γιατί ε, ελέγχει το κατά πόσον είναι απαραίτητη αυτή η έλεγχη, όλα αυτά υποβάλλονται στην κρίση μας, στην αξιολόγησή μας. Και το δεύτερο είναι ότι όταν κάνουμε τη χαρτογράφηση, ανέφερα χθε τα σχετικά, δηλαδή εντοπίζουμε πού ε, εντοπίζεται το ενδιαφέρον των κρατών μελών. Σα έγινε παράδειγμα, βλέπουμε ότι κάποια κράτη ε, οι συγκητές μας το διαπίστωσαν, έχουν ενδιαφέρον για κάτι θέμα. Οι κύριε Κοέλιο και Λόπες Αγγιλάρ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα. Ο κύριο Κοέλιο που ήταν και συγκητής το ΣΕΝΚΑ θα πάρει πρώτο τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νίλσον για την παρουσίαση αυτή εμείς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το Σέγγεν και πώς θα το προστατεύσουμε, ιδίως σε μια πολιτική στιγμή με ε, λαϊκισμού που επιτίθεται κατά της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια συστηματική αξιολόγηση του Σέγγεν για να δούμε πώς τα πηγαίνει, εάν υπάρχουν προβλήματα και πώς θα τα διορθώσουμε. Για αυτά που είπε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τονίσω τα εξής. Πρώτον, έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης. Θα πρέπει εδώ να καταγράψουμε ότι οι έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί από χώρες όπως η Πολωνία, οι κατοχώρες, το Βέλγιο, δείχνουν ότι υπάρχει μία εύλογη χρήση του συστήματος και δεν προκαλούνται προβλήματα. Είναι πιο ανησυχητικό ότι υπάρχουν παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα παρά κάτι άλλο. Οπότε η διαδικασία αξιολόγησης που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιους χώρες θα δώσει ελπίζουμε τα ε, απαραίτητα αποτελέσματα. Με αυτή την ευκαιρία να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι άλλη μια φορά τόνισε ποια ήταν η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Δηλαδή να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια που είναι αδικαιολόγητα και να επιτρέψουμε και στις χώρες αυτές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο χώρο του Σέγγεν. Τρίτον, πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς το νέο σύστημα αξιολόγησης του Σέγγεν. Περιμένουμε την επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε τότε να έχουμε ακόμη περισσότερες και ουσιαστικότερες πληροφορίες για την ε, χρήση του συστήματος. Να θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο ε, σωστά έχει πει ότι η αξιολόγηση του Σέγγεν ε, με χαρακτήρα πιο κοινοτικό είναι μια από τις διαδικασίες που θα προσφέρει περισσότερη αξιοπιστία στο όλο σύστημα, στο χώρο του Σέγγεν. Διότι μόνο με συστηματική αξιολόγηση μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα, ο χώρος Σέγγεν λειτουργεί σωστά. Επίσης, να συγχαρώ σε τέταρτη φάση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που μας είπε, δεν ήταν σαφές αυτής εξ αρχής, ότι οι μη προειδοποιημένες επισκέψεις και εδώ ξέρουμε ότι το Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες στο σύστημα αξιολόγησης του Σέγγεν, ε, μόνον τακτικές. Ε, τέλος πάντων, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλό είναι που οι αποειδοποιητέ επισκέψεις δεν περιορίζονται μόνο στις χώρες που αξιολογηθούν φέτος ειδικώ, αλλά σε οποιοδήποτε κράτος που συμμετέχει στο χώρο του Σέγγεν. Έτσι μπορεί να εντοπιστούν καταστάσεις μη σεβασμού με τους κανόνες του Σέγγεν. Αυτό είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχαίρω και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κάρλος. Thank ε, Χωσέ, ευχαριστώ, Κλοντ. Ενδιαφέρον τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε την έκθεση αυτή αξιολόγησης του Σέγγεν είναι από τα πιο πολύτιμα και ε, αξιόλογα εργαλεία που έχουμε στην ε, προεκλογική εκστρατεία τονίσαμε πολύ από εμά ότι η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι το ευρώ και η εσωτερική αγορά, είναι τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να κινούνται ελεύθερα, να κυκλοφορούν και ε, μας ανάγκασαν όμως επανειλημμένα να θυμίσουμε ότι το Σέγγεν ακριβώς επειδή είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία της όλης ευρωπαϊκής προσπάθειας, δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω, δεν το Σέγγεν κάτι που ταυτίζεται με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μέλη της Ένωσης που δεν είναι στο Σέγγεν, βλέπει Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αντίθετα κάποια κράτη-μέλη που δεν είναι στην Ένωση συμμετέχουν στο Σέγγεν. Αυτό σπανίως το λέμε. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα ζήτημα που εκρεμεί Ρουμανία και Βουλγαρία. Είναι σημαντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και καιρό. Πότε θα δοθεί πλήρες καθεστώς στο Σέγγεν. Δεν υπάρχει ομοφωνία γι' αυτό, δεν τα βρίσκει το Συμβούλιο. Θα πρέπει ακριβώς να κατονομάσουμε ποια κράτη-μέλη αντιδρούν. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν κάνει αυτά που είχαν αναλάβει και δεν είναι απλώς λυπηρό, είναι έσχος που ακόμα δεν ε, έχει εφαρμοστεί αυτό. Το ξέρω ότι είναι θέμα του Συμβουλίου με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή κάποιο σχόλιο σχετικά με τη συμπεριφορά και τη στάση των κρατών μελών που, που είναι μέλη του Σέγγεν χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς πάει εκεί. Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και στα πρότυπα αντίστοιχα με τις χώρες της Ένωσης που δημιούργησαν τη διαδικασία του Σέγγεν. Και είχαμε και ένα επεισόδιο με το δημοψήφισμα στην Ελβετία που γέννησε μια συζήτηση την οποία είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Ήταν μια μονοθεματική συνεδρίαση εδώ της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ρωτώ ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων τώρα, τι μεσολάβησε, ποιε ήταν οι επόμενε εξελίξει και τι περιμένουμε να βγει από αυτό το ελβετικό επεισόδιο, για να το πω έτσι. Ε, και πώς θα επηρεάσει την όλη επίδοση και την αξιολόγηση της λειτουργίας του Σέγγεν. Ο κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ. Uh η εικόνα της κατάστασης σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν που μας δίνει η έκθεση της Επιτροπής αποδεικνύει πόσο μονόπλευρη και άδικη είναι οι κανονισμοί Δουβλίνο 2 και Δουβλίνο 3 σε βάρος των μεσογειακών κρατών μελών. Η Επιτροπή μας ενημερώνει ότι η Κεντρική Μεσόγειος και η Ανατολική Μεσόγειος είναι οι δύο διαδρομές στις οποίες εμφανίζονται οι υψηλότεροι αριθμοί περιπτώσεων παράτυπης διέλευσης των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σέγγεν. Αντίθετα όμως, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό περιπτώσεων παράτυπης διαμονής, τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων είχε η Γερμανία, ακολουθούμενη από τη Σουηδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Η έκθεση παραδέχεται έτσι ρητά ότι το ταξίδι των περισσότερων παράτυπων μεταναστών δεν τελειώνει όταν διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα, αλλά συνεχίζεται με άλλους προορισμούς στον χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, με τους κανονισμούς Δουβλίνο 2 και Δουβλίνο 3, οι συνέπειες του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης επιρρύπτονται κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη από τα οποία γίνεται η αρχική διέλευση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σέγγεν, δηλαδή πρακτικά στην Ιταλία και την Ελλάδα. Έτσι τα κράτη αυτά μετατρέπονται σε ένα είδος αλεξικέραυνου για να προστατευθούν τα κράτη-μέλη της Βόρειας Ευρώπης χωρίς να δίνονται καν τα οικονομικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ώστε τα κράτη πρώτης διέλευσης των συνόρων να μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τόσο απαιτητική αποστολή. Ειδικά μάλιστα για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής και δημοσιονομικής κατάρρευσης, αυτό καταλήγει στο να συσσωρεύονται οι παράτυπα διερχόμενοι μετανάστες που συλλαμβάνονται από τις αρχές σε κέντρα κράτησης κάτω από απάνθρωπες συνθήκες συνοστισμού και εγκλισμού για απαράδεκτα μακρά χρονικά διαστήματα. Αποτελεί συνεπώς επιτακτική αναγκαιότητα η ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος των κανονισμών Δουβλίνο 2 και Δουβλίνο 3 προκειμένου την κύρια ευθύνη για το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης να την αναλάβουν τόσο από οικονομική όσο όμως και από πρακτική άποψη οι χώρες που αποτελούν τον τελικό προορισμό των μεταναστών και όχι οι χώρες διέλευσης. Μόνο έτσι θα βρει έμπρακτη εφαρμογή η αρχή της αλληλεγγύης που κατοχυρώνεται θεωρητικά στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο έτσι οι χώρες τελικού προορισμού θα μπορούσαν να αποδείξουν την προσήλωσή τους στην ιδέα μιας πραγματικά ενωμένης Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σεράια Πολ στην επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Αυτό το οποίο ε, σκεφτόμουν ε, ακούγοντας περί ελεύθερης μετακίνησης είναι ότι είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη όμως όπου η διοίκηση δεν γνωρίζει πώς ε, πρέπει να αντιμετωπίσει τα παρατύπως διερχόμενα άτομα. Για παράδειγμα, στη χώρα μου τη Σουηδία υπάρχουν 800 άτομα που ανήκουν στην κοινότητα των Ρωμά, που ουσιαστικά ε, τους έγινε έξωση από τα σπίτια τους χωρίς κάποια αιτιολογία. Οι δημόσιες αρχές πολύ απλά δεν γνωρίζουν ούτε κατανοούν τα θέματα αυτά. Δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν ακροδεξιές ομάδες στη Σουηδία, οποίες εκμεταλλεύονται και πολύ καλά μάλιστα την κατάσταση. Και βελτιώνουν και τα εκλογικά τους αποτελέσματα ως εκ τούτου. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα ε, τα πράγματα. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη δημοκρατία και πώς μπορεί να ενημερωθούν σωστά τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπληρώνουν το καθήκον τους και πρέπει να ενημερώνουν σωστά τους διοικητικούς φορείς σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ Σωράγια. Η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω μερικές ερωτήσεις αλλά προηγουμένως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ τα θέματα αυτά. Έχω τώρα τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, για τη Frontex. Είπατε ότι 12 είναι τα κράτη που δεν έχουν δώσει ακόμα αριθμητικά στοιχεία για το Frontex και ότι υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που έχουν δώσει πληροφορίες αλλά είναι ελλειπείς. Γιατί παρατηρείτε αυτό, γιατί δεν σας στέλνουν τις πληροφορίες. Είναι προθυμία ή έχουν τεχνικά προβλήματα ή αμέλεια, για ποιο λόγο. Γιατί έτσι δεν ανταποκρίνονται, δεν συνεργάζονται τα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια, βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα με το θέμα αυτό των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όταν φτάνουν αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ένωση, τους παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Αρνούνται τα κράτη-μέλη, το αποφασίζουν τα ίδια, είναι στη διακριτική τους ευχαίρεια, αν θα, πάρουν, αν θα γίνει αυτή η δακτυλοσκόπηση ή όχι μήπως δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση των αστυνομικών ή δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα οι αστυνομικοί και αυτό έχει συνέπειες, ε, κινδύνους. Για ποιο λόγο διαφέρει η αντιμετώπιση. Και τι ε, συνέπειες έχει αυτό για τις αιτήσει ασύλου. Αλλάζει η διαδικασία ανάλογα αν έχεις δώσει ή δεν έχεις δώσει τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Επιταχύνονται, επιβραδύνονται. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγα περισσότερα σχετικά. Και επίσης είδα κάποιες ελλείψεις και κάποιες αδυναμίες τους μηχανισμούς αξιολόγησης της λειτουργίας του Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς σκέφτεται να το αντιμετωπίσει αυτό και να αντιδράσει. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τελευταία ομιλήτρια κυρία Winberg. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι κάτι που αφορά ιδιαίτερα και τη Σουηδία πολλοί έχουν καταλήξει να θεωρούν το θέμα αυτό συνοψίζεται στο να ξεφορτωθούμε τους μετανάστες από τη Ρουμανία. Αλλά τελικά προσφέρουμε και ένα ταξίδι δωρεάν για επιστροφή στη Ρουμανία. Ε, αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι η Ρουμανία θα πρέπει να ασχοληθεί με την ένταξη τώρα Ρωμά στην ε, ίδια τη Ρουμανία και να ασχοληθεί με τους πολιτές της χώρας της. Ο Ρουμάνος πρέσβης έχει ε, ήδη τοποθετηθεί για το θέμα της ε, επαιτίας στη Σουηδία, με το οποίο έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πραγματικά πολλές δυσάρεστες καταστάσεις που δημιουργούνται σε σχέση με αυτού του είδους τα φαινόμενα και τη μετανάστευση και πραγματικά η Ρουμανία θα πρέπει να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση που ήδη λαμβάνει ώστε να φροντίσει για την ένταξη του δικού της πληθυσμού Ρωμά. Εάν δει κανεί τι συμβαίνει και με το δίκτυο Eurodac και τα σχετικά ζητήματα, όταν κανεί ε, παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα, Η περίοδος, τήρησης, η περίοδος τήρησης των δεδομένων είναι 18 μήνες. Μετά ε, η βάση δεδομένων ε, αδειάζει. Και είναι και πολλά τα κάτι μέλη που δεν παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τον αριθμό των ανθρώπων και την εισρωή μεταναστών. Ε, θα θέλαμε και ως προς αυτά λοιπόν κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο λόγος πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλα τα θετικά σχόλια σε σχέση με την έκθεση. Θα σταθώ σε κάποια σημεία. Πρώτα απ' όλα, όντω, όπω είπε ο κύριο Κουέλιου, ο νέο μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν, αυτό καθεαυτό, το μέλλον, θα είναι μια βασική πηγή άντλησης πληροφοριών και δεδομένων για τέτοιου είδους εκθέσεις. Οπότε θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε κάπως καλύτερα μόλις έχουμε τα πρώτα πορίσματα από την λειτουργία του νέου μηχανισμού ε, να είναι εκθέσεις πληρέστερες και διεξοδικότερες για το πώς λειτουργεί ο χώρος Αυτή είναι και η πρόθεσή μας. Για τι συνδυόμενε χώρε δεν μπορώ να πω εάν τα έχουν πάει καλύτερα ή χειρότερα από οποιοδήποτε κράτο μέλο ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση με το κεκτημένο Σέγγεν. Έχουμε κάποια παράπονα και κάποιε ε, αιτιάσει κατά των χωρών αυτών, όπω όμω και με τα κάτι μέλη του χώρου Σέγγεν, αλλά δεν υπάρχει λόγο να σταθούμε ιδιαίτερα στη σκοπιά τη ε, συμμόρφωση με το κεκτημένο το δημοψήφισμα στην Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία από νομικής ε, άποψης και μόνο ε, δεν αφορά την ε, συμφωνία Σέγγεν άμεσα. Είναι δύο ανεξάρτητες συμφωνίες. Όμως ανάλογα με το τι θα σκεφτεί και τι θα αποφασίσει να κάνει η Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να υπάρξουν συνέπειες και για το Σέγγεν και βεβαίως θα υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων του τομέα. Για τα υπόλοιπα σχόλια δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω απηχούν ε, το εξής βασικό ζήτημα. Το Σέγγεν είναι περίπλοκος προς την ε, παρακολούθησή του και το, το να γνωρίζει κανείς το αν λειτουργεί καλά υπάρχει ε, και άμεση συνέπεια με το τι θα γίνει με το Σέγγεν, με το Σέγγεν γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα όπως ε, για το άσυλο, για τους εκόντες άσυλο ή για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων. Αυτά όλα σχετίζονται με την ε, υλοποίηση του κεκτημένου Σέγγεν. Είναι λοιπόν περίπλοκο το σύστημα από μόνο του σε ό,τι αφορά την συλλογή δεδομένων Frontex και γιατί τόσα πολλά κράτη-μέλη δεν ε, προσφέρουν τις ε, απαιτούμενες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση αυτή η όλη διαδικασία είναι καινούρια. Η Frontex ε, άρχισε να ζητά δεδομένα από τα κράτη-μέλη, κάποιοι καθυστέρησαν ή τα έστειλαν. Ίσως να είναι δύσκολο να τα καλύψουν όλα αυτά τα κατι μελη και να τα συγκεντρώνουν συστηματικά. Και μάλιστα το θέμα δεν είναι να καταγράφει κανεί μόνο το ποιοι συλλαμβάνονται στην επικρατεία ενό μέλου ω παρανόμω διαμένοντε, αλλά και να γνωρίζει την, τον τόπο προέλευση και το πώ έφτασαν ω εκεί. Ε, είναι διαφορετικά αυτά όμως που θα ενδιαφέρουν κάποιον που ασχολείται με θέματα ασύλου. Ε, να σας δώσω τώρα ένα υποθετικό κλασικό παράδειγμα. Κάποιος φτάνει στη Γερμανία ε, αεροπορικός. Το θέμα είναι να δει λοιπόν αν πέρασε κανείς αυτός που συλλαμβάνει εκεί μόνο για να πάει αλλού ή αν έχει σκοπό να παραμείνει στη Γερμανία ή να αιτηθεί άσυλο. Εδώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει πιο συστηματικά να συλλέγουν λοιπόν τα δεδομένα, να τα στέλνουν στη Frontex σίγουρα, αλλά είναι δύσκολο να το κάνουν όλοι την ίδια στιγμή. Θα γίνει, αλλά θα καθυστερήσει. Και εφόσον συλλέγουμε και τα δεμένα αυτά, θα δούμε πώ λειτουργεί το Σέγγεν και ω προ αυτή τη διάσταση. Κάποιε παρατηρήσει τώρα για τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα παρακολουθούμε αυτά τώρα. Είδαμε να υπάρχουν κάποια παράπονα κάτι κράτη-μέλη με κάποιους ε, που έχουν εντοπιστεί, συλληφθεί, να λένε ότι μπήκαν στο χώρο Σέγγεν από άλλο κράτος μέλος που όμως δεν ε, έκανε, δεν ανέλαβε τις, και δεν υλο, εφάρμοζε τις διαδικασίες που προβλεπόνται με το σύστημα Eurodac. Δεν ε, συμμορφώνονται λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε και τους λόγους. Κάποιες φορές οι μετανάστες απλώς αρνούνται να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Τώρα, τι μέτρα καταστολής μπορεί κανείς να προβλέψει τότε, τι είναι νομικός, αποδεκτό, αναλογικό, υπάρχει πρόβλημα συμμόρφωσης των κρατών μελών, με τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή, αλλά το συζητάμε ακόμη με τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι κάλυψα τα βασικά ζητήματα με αυτές τις παρατηρήσεις. Εάν κάτι ξέχασα, πείτε το μου. Πριν φύγετε, ε, θα ήθελα να πω από πλευράς του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Αφιερώνουμε πολύ χρόνο και ενέργεια στην ε, μεταρρύθμιση της ε, διαχείρισης του Σέγγεν και της αξιολόγησης και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και τις εθνικές αξιολογήσεις και θα κάνουμε και πρόταση μετά τις θερινές διακοπές. Ε, πολύ καλή συζήτηση ήταν και οι συνάδελφοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το Σέγγεν γιατί θα καταλάβετε ότι είναι πολύ περισσότερα από την ελεύθερη κυκλοφορία και τα θέματα ασφαλείας είναι και θεωρήσεις διαβατηρίων, εξασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα επανέλθουμε βέβαια με την πρόταση και θα αναπτύξουμε αυτή τη συζήτηση σε λεπτομέρειες μετά τις τελευταίες διακοπές. Λοιπόν, μιλήσατε όλοι πολύ ειλικρινά και πολύ ελεύθερα και επιτηρήσατε και το χρόνο αγόρευση. Ελπίζω να μην κουραστήκατε, γιατί έτσι θα πάει ο ρυθμός και μετά το καλοκαίρι. Και το λέω στους νέους βουλευτές, συνεχίστε να είστε τόσο επιμελείς. Και ελπίζω να μην ε, σας ε, σταματώ. Δεν τελειώσαμε. Θα έρθει και η νομική υπηρεσία. Με διακόπτη γραμματεία. Τι έχασα και τον ήρμό τώρα. Συγγνώμη. Δεν λέω να φύγουμε. Ε, δεν, δεν κλείνω τώρα. Έχουμε και άλλο θέμα. Απλώ λέω να συνεχίσουμε έτσι αυτή την παρουσία και την ε, τακτική στι συνεδριάσει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και έτσι θα πάει και μετά το καλοκαίρι. Λοιπόν, αν θέλετε να παραμείνετε για το επόμενο θέμα. Μπορεί να φαίνεται άχαρο και διεκπαιρεωτικό, αλλά είναι ενδιαφέρον. Είναι παρουσίαση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Ο τίτλος μόνο είναι τόσο μακρύς. Βασικά πρόκειται ε, για την πειρατεία. Θα δώσω αμέσω το λόγο στη νομική υπηρεσία. Ποιος είναι εδώ από την νομική υπηρεσία, ο κύριος Άλεκ. Ζητώ συγγνώμη που σας δίνω το λόγο έτσι με τέτοιο στενό, στεγνό τρόπο αλλά κάναμε τέτοια ωραία συζήτηση, τόσο ενδιαφέρουσα και ήθελα να συνεχιστεί και τώρα πάμε σε αυτά τα στεγνά και άχαρα θέματα τα νομικά. Είναι πολύ σημαντικό όμως. Ε, και η νομική υπηρεσία λίμωνο για μας μας βοηθάει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ να σας ενημερώσω για την ε, υπόθεση που ξεκίνησε το δικαστήριο πριν από τρία χρόνια μετά από δική σας πρωτοβουλία Λίβε, μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών και πρόκειται ακριβώς για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για τους όρους της μεταγωγής των υπόπτων πειρατείας και των συναφών κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από ε, τις ε, δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού ε, στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Μαυρικίου. Ήταν μια συμφωνία που έγινε στα πλαίσια της στρατιωτικής συνεργασίας Αταλάντη, αν θυμάστε τότε, στον κόλπο του Άντεν κατά της πειρατείας. Στις 24 Ιουνίου φέτος το ΔΕΚ διατήρησε την ε, προσφυγή του Κοινοβουλίου και αποφάσισε να ακυρώσει την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Ιουλίου 2011. Ποια είναι τα προβλήματα και γιατί ελήφθη μια τέτοια απόφαση τελικά. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι το Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή τη συμφωνία μετά ε, αποκλειστική ε, βάση το άρθρο 37 που είναι για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Δηλαδή το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε καθόλου ούτε στη διαδικασία διαβούλευσης ούτε στην καταληκτική ούτε ζητήθηκε σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, ούτε τίποτα. Ήταν όλα ερήμη του Κοινοβουλίου, ούτε καν ενημερώθηκε. Ε, προσφύγαμε στο δικαστήριο και ε, έχουμε δύο καινοτομίες από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Πρώτον, ε, η ρήτρα αποκλειστικότητας, το άρθρο 286, 218.6, όπου το Συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία ε, χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά μόνο σε τομείς ΕΠΑΑ. Ε, και επίσης ζητήσαμε την ερμηνεία του Κοινοβουλίου για το δικαίωμα πληροφόρησης του Κοινοβουλίου ε, στο άρθρο 218 παράγραφος 20. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ασμένος και πλήρως να ενημερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια και τις φάσεις από την αρχή μέχρι τη σύναψη της τελικής συμφωνίας. Όταν λοιπόν αναλύσαμε τους στόχους και το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής με το Μαυρίκιο, διαπιστώσαμε ότι δεν καλύπτει μόνο ε, πτυχές εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, αλλά και δικαστική συνεργασία στο ποινικό δίκαιο ε, για την δικαιοδοσία ε, των δικαστηρίων του Μαυρικίου, η αστυνομική συνεργασία, συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών, καθώς επίσης και αναπτυξιακή συνεργασία, γιατί η ίδια η συμφωνία αφορά αναπτυξιακή βοήθεια προς το Μαυρίκιο. Άρα δεν ήταν μόνο και μάλιστα ε, και με γραμμές ε, από τον προπολογισμό της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Για πρώτη φορά αποφάνθηκε το δικαστήριο για τη ρήτρα αποκλειστικότητας και ότι η συνθήκη της Αφώνας μπορεί να βρει διάφορες ερμηνείες. Υποστήριξε το δικαστήριο την εσωτερικό καταμερισμό εξουσιών και και τη νομική βάση, οπότε θεώρησε ότι θα πρέπει να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου εάν ε, ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι εκτός της ε, ΕΠΑ. Άρα εδώ στη συμφωνία υπάρχουν διάφοροι στόχοι χωρίς να επικυριαρχεί κανένας επί των άλλων. Σήμερα θα επικεντρωθώ στο, στη δεύτερη ε, αξίωση της ΛΥΜΠΕ για το πώς ε, ε, ερμηνεύει το δικαστήριο το άρθρο 218-20. Το Συμβούλιο ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι αρχίζουν διαπραγματεύσεις το Μάρτιο του 2010. Και την επόμενη φορά που έμαθε οτιδήποτε το Κοινοβούλιο για τη συμφωνία αυτή ήταν τον Οκτώβριο του 2011. Τρεις μήνες μετά την υπογραφή και την ολοκλήρωση και τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Ε, και αφού είχε ε, δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα. Δηλαδή ήταν ε, σε πλήρη άγνοια των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο, γιατί έτσι το κρατούσε το Συμβούλιο απομονωμένο. Και εδώ το δικαστήριο έλαβε θέση σαφή ότι αυτό ήταν παραβίαση της βασικής διαδικασίας και των απαιτήσεων αυτής στην απόφαση του Συμβουλίου. Οπότε ακύρωσε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου κανονικά. Τώρα, τι μπορούμε εμείς να εξαγάγουμε ως συμπέρασμα. Είπε ξεκάθαρα το άρθρο ότι το 2.18.10 της συνθήκης είναι δεσμευτική ρύθμιση και όχι απλή ε, διακήρυξη. Και ο στόχος είναι να βεβαιωθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να ασκεί το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο στην ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και να κάνει τη φωνή του να ακούγεται και τις απόψεις του σεβαστές. Έτσι εκφράζονται οι δημοκρατικές αρχές στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια το δικαστήριο είπε ξεκάθαρα ότι ε, εφόσον έχει παραβιάσει αυτά το Συμβούλιο ε, κηρύσσεται άκυρη η απόφαση του και αυτό είναι ε, στην πλήρη δικαιοδοσία του ΔΕΚ. Το άρθρο 218 καλύπτει κάθε είδους ε, συμφωνίες, συμφωνίες ε, που εμπίπτουν στη δική σας αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ, που δεν είναι αποκλειστικά της εξωτερικής πολιτικής. Και επίσης είπε το δικαστήριο ότι αφορά όλες τις φάσεις, από την αρχή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις οδηγίες για τη διαπραγμάτευση, η όλη διαπραγμάτευση, η μονογραφή, η υπογραφή, ε, τα συμπεράσματα και ε, η επόμενη φάση που μπορεί να είναι η αναστολή ε, ή η διακοπή της εφαρμογής και θα πρέπει πάντα να είναι πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο. Βέβαια αυτά όλα τα λέει το δικαστήριο. Το Κοινοβούλιο τώρα πώς μπορεί να βασιστεί και να προχωρήσει και τι επιπτώσεις θα έχει για την Επιτροπή σας αυτό. Πρώτον, μία εκδοχή είναι στις ακροάσεις των Επιτρόπων να το συζητήσετε με το νέο υποψήφιο ορισμένο Επίτροπο για το πώς προτίθεται να εφαρμόσει αυτή την απόφαση του δικαστηρίου και πώς θα γίνει αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Διοργανική Συμφωνία. Δεύτερον, βεβαίως η απόφαση δίνει κάθε δικαίωμα στο Κοινοβούλιο να εκφράζει την άποψή του στις διαπραγματεύσεις και το συνδέει με το δημοκρατικό έλεγχο και αυτό αφορά και την ουσία και τον τύπο της ε, διαδικασίας και της διαπραγμάτευσης το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πλήρως προς το σκοπό αυτό να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο μπορεί πάντα να ρωτάει ε, πώς λαμβάνονται υπόψη οι θέσει του και πώς συμπεριλαμβάνονται στην ε, συμφωνία και την τελική αξιολόγηση. Είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να εκφράζει την άποψή του το Κοινοβούλιο για αν θέλουμε μια προσωρινή ε, εφαρμογή πριν δώσει το Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του και τεθεί σε και όταν όλα αυτά δεν τηρούνται και υπάρχει βασική παραβίαση θα ε, έχει την πλήρη δικαιοδοσία το δικαστήριο να αποφασίσει. Τέλος, έχουμε μια δεύτερη αντίστοιχη ε, περίπτωση υπόθεση στο δικαστήριο κατά της απόφασης του Συμβουλίου για αντίστοιχη ε, συμφωνία με την ε, Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, πάλι για τους πειρατές, το ίδιο θέμα, όχι το Μαυρίκιο. Και πάλι ούτε καν ενημερώθηκε το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος πολύ πιο γρήγορα και δεν θέλω να σα πιέσω, αλλά ήταν όλοι πολύ σύντομοι και τα καταφέραμε πολύ γρήγορα. Όλοι θέλουν να προλάβουν και να πάνε διακοπέ γρηγορότερα. Σε κάθε περίπτωση, στην νομική υπηρεσία να πω ότι είσαστε πολύτιμοι για μα, παρόλο που σα πιέσαμε λίγο για να βιαστούμε και είναι πολύ σημαντική η απόφαση αυτή για τη λειτουργία τη Επιτροπής μα διότι παρακολουθούμε το πώ διαμορφώνονται πολλέ διεθνεί συμφωνίε. Ε, πρέπει να υπάρχει το επαρκές επίπεδο πληροφόρησης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, βελτιώνουν διαρκώς τις σχετικές διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τις ακροάσεις της Επιτροπής να τις παρακολουθούμε διότι είναι πολλά τα στοιχεία που μας δώσατε και είναι και πολλές και οι συνέπειες που θα υπάρξουν για μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερως για αυτήν την ε, παρουσίαση. Με αυτά τα λόγια νομίζω πραγματικά πολύ νωρίτερα μπορούμε να φτάσουμε στις ευχαριστίες μου προς τα μέλη, να σας ευχηθώ καλές διακοπές, το ίδιο και σε όλους ε, τους εργαζομένους στην Επιτροπή μας. Καλές σας διακοπές και θα σας ξαναδούμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε.